Good day. Bonjour à tous. Buenos días. Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλημέρα σας. Παρακαλώ καθίστε. We should be ready to kick off and get going. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Στη δημόσια μας ακρόαση για το πώς θα ξεμπλοκάρουμε την οδηγία κατά των διακρίσεων. Εκρεμεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, και για την δική μας Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για οδηγία που εφαρμόζει η συμμεταχείριση μεταξύ των ανθρώπων ανεξάρτητα της θρησκείας, ηλικίας, πίστης ή γενετήσιου προσανατολισμού. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδοκίμασε την πρόταση και η συγγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν η Καθλίν Μπέιτενβεχ. Και μάλιστα υιοθετήσαμε και μια γνωμοδότηση με βάση τη διαδικασία διαβουλεύσεων στις 2 Απριλίου του 2009 και μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας το Δεκέμβριο του 2009 η πρόταση πια αυτή εμπίπτει στο άρθρο 19 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται ομοφωνία από το Συμβούλιο και συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα έχουμε ορίσει ένα νέο εισηγητή για το θέμα αυτό, τον συνάδελφό μας ε, Ραούλ Ρομέβα, η Ρουέδα, και εξετάσαμε τη μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έδειξε ότι ενώ η έλλειψη διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πράξη το επίπεδο νομικής προστασίας για την εξασφάλιση του σεβασμού αυτής της αρχής ε, ε, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Οπότε το θέμα αυτό έχει κολλήσει τα τελευταία χρόνια στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης στο Συμβούλιο. Και δεν είναι καθόλου ευνηδιαστικό, δεν είναι ε, η μόνη περίπτωση που έχουμε έναν ευαίσθητο, έναν ευαίσθητο δοσιέ να μπλοκάρεται στο Συμβούλιο παρά τις ε, άοκνες προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προωθήσει το θέμα. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επανειλημμένος ε, και εντόνως να συνεχιστούν οι συζητήσεις και να προωθηθεί το θέμα, δυστυχώς ε, ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής. Γι' αυτό και οργανώνουμε αυτή τη δημόσια κρόση προκειμένου να δώσουμε μια νέα όθηση και να βοηθήσουμε και εμπράκτος ε, στην απεμπλοκή αυτού του θέματος, αυτής της οδηγίας δηλαδή κατά των διακρίσεων. Η συζήτησή μας και η ακρόασή μας χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα επικεντρώνεται στα θεσμικά ζητήματα και θα ακούσουμε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή την πορεία των διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά την οδηγία κατά των διακρίσεων. Θα έχουμε εδώ στο πρώτο τμήμα τον κύριο Τσοβάνο Τορντέα που είναι ο Διευθυντής ε, Ισότητας και Δικαιοσύνης στην Αρμόδια Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλώς ήρθατε κυρία Ντορντέα και την κυρία Χεσελέγκερ που εκπροσωπεί το Δανικό Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης. Εκπροσωπεί την Δανική Προεδρία. Και σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε στην ε, δημόσια αυτή ακρόαση. Μετά το πρώτο τμήμα θα έχουμε δύο ακόμη τμήματα στη δημόσια ακρόαση. Εκεί θα κάνουμε μια επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου ε, ίσης μεταχείρισης και ε, κατάργησης των ε, διακρίσεων και θα δούμε τους λόγους ε, διακρίσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 19 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δούμε ποιε θα πρέπει να είναι οι βασικές αρχές μιας ε, περιεκτικής οδηγίας κατά των διακρίσεων. Μετά το δεύτερο τμήμα θα έχουμε ένα γύρο ερωταπαντήσεων μεταξύ των μελών και των ε, προσκεκλημένων του πάνελ, οπότε ετοιμάστε ήδη τις ερωτήσεις σα. Και θα έχουμε και ένα τρίτο τμήμα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη δημόσια κρόση με την εισαγωγή του εισηγητού μας, του κυρίου Ρωμέβα Ιρουέδα, και μετά θα ακούσουμε τους δύο πρώτους προσκεκλημένους. Πρώτα λοιπόν ο εισηγητής μας ο κύριος Ρωμέβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την διοργάνωση της αυτή, αυτής της δημόσιας ακρόσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και πολύ φοβούμαι ότι δεν θα είναι ούτε και η τελευταία. Η εισήγησή μου θα είναι αρκετά σύντομη κυρίως γιατί δεν έχω και πολλά να προσθέσω σε αυτά που είπαμε, θα έλεγα τους τελευταίους μήνες, αλλά μάλλον τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία αυτή. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω όμως μερικά στοιχεία που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά για να δούμε πού βρισκόμαστε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ που βρισκόμαστε. Είναι σε αυτή τη στιγμή η έλλειψη βούλησης μελών του Συμβουλίου να απεμπλέξουν ε, μια οδηγία που είναι θεμελιώδη σημασία για τα βασικά δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Πολλοί συμπολίτες μας δυστυχώς δεν καλύπτονται από την νομοθεσία για ορισμένες περιστάσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Κατά τη γνώμη μου, κάτι τέτοιο αντιβαίνει στι ίδιε τι θεμελιώδει αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει οπωσδήποτε να διευθετηθεί. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο είναι τόσο σημαντική αυτή η οδηγία και γι' αυτό επιμένει τόσο έντονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην απεμπλοκή τη κατάσταση. Εμεί εκπροσωπούμε του πολίτε τη Ευρώπη. Οπότε είναι και χρέο και βασικό καθήκον και ευθύνη μα να διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα και να καλύψουμε αυτό το κενό στην ε, κοινοτική νομοθεσία. Ένα άλλο σημείο που είναι πολύ σημαντικό αφορά μια αντίφαση. Εμείς διαπιστώνουμε ότι μερικές χώρες μέλη έχουν νομοθεσία που θα την επιθυμούσαμε και πανευρωπαϊκά και αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια κοινότητα που θέλουμε οι πολίτες μας να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις φυσικά, αλλά κυρίως και τα ίδια δικαιώματα, είναι αδιανόητο που μόνο ο, μερικά κρατημέλη καλύπτουν και σέβονται αυτά τα δικαιώματα, ενώ τα υπόλοιπα κρατημέλη δεν τα εξασφαλίζουν. Γιατί έτσι δημιουργούνται διακρίσει σε ό,τι αφορά την ελευθερία τη διακίνηση των κρατών μελών από τη μία χώρα στην άλλη. Κάτι που αντιβαίνει, επαναλαμβάνω, στι θεμελιώδει αρχέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ζητούμε από όλους τους ε, υπεύθυνου, από όλα τα θεσμικά όργανα και τους ηθήνοντες να σβρώξουν τα πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση και να, ξεμπλέ, ξεμπλέξουμε από αυτό το αδιέξοδο. Όπως μας είπε και ο Πρόεδρος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, υπερψήφισε μια γνωμοδότηση το 2009, τον Απρίλιο του 2009. Το ψήφισμα αυτό δίνει ένα ηχηρό μήνυμα και οθεί τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήταν πολύ δύσκολη η επίτευξη συνένεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και ήταν πολύ καλό το ψήφισμά μας με εισηγήτρια την κυρία Κατλίν Μπέιτεμβεχ. Και αυτή είναι η βάση του σημείου αφετηρίας και για τη σημερινή μας θέση. Θα ήθελα να πω ότι κάτι είναι πολύ σημαντικό όταν προσεγγίζουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι ότι μιλούμε για ένα πακέτο δεν θα πρέπει να κατακαιρματίζουμε το πακέτο σε επιμέρους σημεία. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως σύνολο. Να καλύψουμε ό,τι δεν καλύπτεται και δεν μπορούμε να αρχίσουμε τα παζαρέματα για το τι μας ενδιαφέρει περισσότερο, τι είναι πιο σημαντικό και τι άλλο. Όλα είναι σημαντικά, το σύνολο του πακέτου είναι σημαντικό. Δεν θα πρέπει να το διαιρέσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σύνολο. Δεύτερον, κάποια από τα επιχειρήματα που ακούσαμε στο πρόσφατο παρελθόν και που συνδέονται με την ε, σοβούσα οικονομική κρίση είναι ένα παραπέτασμα καπνού ουσιαστικά. Κάτι που προσπαθεί να συγκαλύψει το ουσιαστικό πρόβλημα που είναι η έλλειψη βούλησης κάποιων μελών του Συμβουλίου να συμφωνήσουν με την ε, νομοθεσία αυτή κατά των διακρίσεων. Αυτό θέλουμε λοιπόν, ένα ηχηρό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ξεμπλέξουμε τις συζητήσεις για την οδηγία αυτή. Εγώ συγητής ε, πρότεινα τη διοργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόαση γιατί παρακολούθησα το έργο των τελευταίων προεδριών και διαπίστωσα ένα τρομερό πρόβλημα. Αρχίσαμε την κοινοβουλευτική μας θητεία, την τελευταία, με την Ισπανική Προεδρία. Ε, η ισπανική δυσκολία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, με πολύ θαραλέο τρόπο έθεσε το ζήτημα επιτάπητος και προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα διάφορα πρακτικά προβλήματα. Στη συνέχεια είχαμε τη Βελική Προεδρία, μετά την Ουγγρική, αλλά ε, διαπιστώσαμε μια αποδυνάμωση της βούλησης της Προεδρίας να προωθήσει το θέμα. Εγώ σας ε, ομολογώ ότι έχω υψηλέ προσδοκίες από την Δανική Προεδρία. Γι' αυτό και επανέφερα το θέμα στην Δανική Προεδρία, γιατί η Δανία έχει δεδηλωμένη ε, δέσμευση και προσήλωση στα θέματα αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό για να προταστατήσει η Δανική Προεδρία στη συζήτηση. Το ζητούμενο από την ακρόαση είναι να βοηθήσουμε τη Δανική Προεδρία να κρατήσει ζωντανό αυτό το θέμα, να το κρατήσει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και να μην το αρχιοθετήσει. Να το θέσει ενώπιον των κρατών μελών ζητώντας μία πρόοδο των συζητήσεων. Νομίζω ότι είναι σημαντική ανάγκη αυτή της ευρωπαϊκής κοινωνίας και σημαντική προσδοκία των Ευρωπαίων πολιτών. Εδώ έχουμε δύο μέτωπα στα οποία μπορούμε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Το ένα είναι απέναντι στην Κομισιόν και το άλλο απέναντι στο Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω δύο ερωτήσεις προς τα θεσμικά όργανα και μετά κατά τέλος των εισηγήσεων θα έχουμε και ερωταπαντήσει. Θα ήθελα να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το μέχρι τώρα έργο της και είναι σημαντικό να συνεχιστεί αμύωτη αυτή η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει την απεμπλοκή της κατάστασης στο Συμβούλιο τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έργο αυτό. Ποιε είναι οι προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τη στάση του προκειμένου να προωθηθεί το ζήτημα. Προς το Συμβούλιο θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για την σημερινή παρουσία της Προεδρίας, γιατί όντως η Προεδρία, η κάθε Προεδρία συνοδεύεται ε, μια, από μια πληθώρα υποχρεώσεων και το ότι βρήκε χρόνο το Συμβούλιο να έρθει εδώ είναι πολύ σημαντικό. Γνωρίζω ότι είναι κάποια κρατημέλη αυτά που μπλοκάρουν την οδηγία. Πάντως, ε, μέλημα του, των εκπροσώπων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διορθώσει αυτή την αδιαφάνεια που επικρατεί στο θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διαφάνεια και η εντιμότητα από όλες τις πλευρές. Θα μας πούν ξεκάθαρα τα κρατημέλη, δεν μας αρέσει αυτό και το α, το β, το γ σημείο. Για να γνωρίζουν όλοι καθαρά και ξάστερα γιατί ορισμένες χώρες ε, αντιστέκονται σε μερικά θεμελιώδη ζητήματα της κοινοτικής νομοθεσίας θα πρέπει με ειλικρίνεια και ετοιμότητα να πούν αυτές οι χώρες τους συμπολίτε τους γιατί τους στερούν δικαιώματα που απολαμβάνουν άλλοι πολίτες σε άλλα κράτη-μέλη. Γιατί εμποδίζοντας τους πολίτες ενός κράτους να έχουν ε, τα δικαιώματα αυτά ε, σε άλλο κράτος, ε, δημιουργεί αντιφάσεις και διαφορές. Αυτές οι αντιφάσεις θα πρέπει να εντοπιστούν και να συζητηθούν. Η πρότασή μου λοιπόν προς το Συμβούλιο και απευθύνομαι εδώ στη Δανική Προεδρία γιατί γνωρίζω την ευαισθησία της για το θέμα αυτό. Ε, και να ρωτήσω τη Δανική Προεδρία πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να απεμπλέξει αυτό το ζήτημα. Αυτά είναι οι εισαγωγής και φυσικά θα υποβληθούν και πολλές τεχνικές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή μας. Τον κύριο Ρωμέβα που <coughs> μας παρουσίασε το θέμα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν κατευθείαν. Στην πρώτη συζήτηση που έχει να κάνει με την θεσμική άποψη. Θα ακούσουμε πρώτα τον ε, κύριο Αουρέλ ε, Τσομπάνου Ντορτέα που είναι ε, Διευθυντής Ισότητας της Γενικής Διεύθυνσης για τη Δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, κύριε Ντορντέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή που οργάνωσε αυτήν τη συζήτηση. Ευχαριστώ και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που ε, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό ε, απέναντι στην ε, κατάσταση και ε, την περίπτωση αυτής της οδηγίας. Είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε τη συζήτηση αυτή και να ακούσουμε όχι μόνο τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία, αλλά να ακούσουμε και τους ενδιαφερομένους, τους εκπροσώπους των πολιτών, σχετικά με τους ε, βαθύτερους στόχους αυτής της νομοθετικής πρότασης. Θέλουμε να ακούσουμε τους πραγματικούς λόγους που χρειάζεται να προχωρήσει στο Συμβούλιο αυτή η νομοθετική πρόταση και που πρέπει να υιοθετηθεί. Επιτρέψτε μου να πάω λίγο πίσω στο 2008 στου ε, στους λόγους που οδήγησαν την ε, Επιτροπή να υποβάλει αυτή την νομοθετική πρόταση έχοντας ε, κατά νου την ανάγκη να γεμίσει ένα, νομικό, ένα νομοθετικό κενό. Ε, είχαμε την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, κατά των διακρίσεων λόγω φύλου, φιλής ή θρησκείας. Αυτά ισχύουν στον τομέα της απασχόλησης και αλλού αλλά ε, οι διακρίσεις ε, λόγω ε, σεξουαλικών προτιμήσεων θρησκείας και αναπηρίες ισχύουν μόνο στον τομέα της εργασίας. Ήδη ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε το θέμα αυτό. Ε, μιλάμε για την νομική προστασία κατά των διακρίσεων που θα πρέπει να παρέχεται στους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα όχι μόνο τους πολίτες αλλά όλους τους ε, ανθρώπους που κατοικούν στο έδαφος των κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν κοινού στόχους όταν μιλάμε για την ε, νομοθετική αυτή πρόταση. Είχαμε κατά νου την ανάγκη να παρέχεται ε, νομική προστασία κατά των διακρίσεων σε τομείς όπου εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, όπου φορείς ισότητας από τα κράτη-μέλη, μέλη του Κοινοβουλίου έχουν λάβει παράπονα. Για παράδειγμα, ε, διακρίσεις εις βάρος ε, μουσουλμάνων σε ξενοδοχείο, παρενόχληση μουσουλμάνων φοιτητών ε, σε, σε φοιτητών σε σχολεία κλπ. μιλάμε λοιπόν για τις πραγματικές ανάγκες πραγματικών ανθρώπων έξω από τα πλαίσια των θεσμικών μας οργάνων. Υπάρχει η ανάγκη προστασίας των ανθρώπων ε, με αναπηρίες ε, και η δυνατότητα να ε, καλύπτονται οι ανάγκες τους με ε, ανάλογες προσαρμογές. Αυτά δεν είναι νέα. Ε, αυτά ήδη έχουν συζητηθεί κατά την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρίες. Και τρίτος σημαντικός ε, στόχος έχει να κάνει με την νομική προστασία ατόμων για με, βάση τις εμπειρίες των κρατών μελών στον τομέα αυτών. Ε, κάτι που ξεπερνάει τα όρια των υπαρχουσών ε, οδηγιών. Ε, και μιλάμε για περιπτώσεις όπου ξεπερνάμε τα όρια της απασχόλησης. Έχουμε πολλά παραδείγματα τα περισσότερα προέρχονται από κράτη-μέλη που στηρίζουν την νομοθετική αυτή πρόταση, καθώς και από κράτη-μέλη που είναι κατά της νομοθετικής αυτής πρότασης, από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Σουηδία, αλλά και από τη Γερμανία. Παραμένουμε πεπισμένοι ότι χρειαζόμαστε την οδηγία αυτή για να ολοκληρώσουμε την προστασία κατά των διακρίσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διακρίσεις ε, λόγω θρησκείας, ε, σεξουαλικών γενετήσεων προσανατολισμού ηλικία και αναπηριών ε, δεν ε, είναι κάτι που μπορούμε να δεχτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ε, στις αρχές του 21ου αιώνα και θα πρέπει η προστασία αυτή να ξεπερνάει τα όρια της ε, αγοράς εργασίας. Ε, έχουμε συλλέξει καλές εμπειρίες ε, με την οδηγία ισότητας λόγω καταγωγής, λόγω εθνοτικής προέλευσης και θέλουμε τις εμπειρίες αυτές να τις ε, εκμεταλλευτούμε και δεν καταλαβαίνουμε γιατί η νομοθετική αυτή πρόταση θα πρέπει να ακολουθήσει άλλη κατεύθυνση από τα θετικά παραδείγματα που είχαμε στο παρελθόν. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Εάν ε, δεν ήταν ε, σαφές αυτό από την επανέμβαση του κυρίου Ρωμέβα. Όλοι γνωρίζουμε ότι ε, το παρόν μπλοκάρισμα της ε, νομοθετικής πρότασης οφείλεται στην ε, πολιτική αντίθεση λίγων κρατών μελών, πολύ λίγων κρατών μελών. Υπάρχει γενική υποστήριξη, τα περισσότερα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο στηρίζουν την νομοθετική αυτή πρόταση, αλλά... Οι συνθήκες προβλέπουν ομοφωνία στο Συμβούλιο για να υιοθετηθεί μια τέτοια πρόταση. Δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν μέχρι τώρα να έχουμε πολιτικό διάλογο με την ε, μειονότητα που αντιστέκεται και η Κομισιόν ε, προσπάθησε κατά τα τελευταία χρόνια με τις ε, διάφορες προεδρίες ε, να ακολουθήσει άλλο μονοπάτι και να καλύψει κάποιες, κάποια από τα σημαντικά πολιτικά θέματα, πολιτικά επιχειρήματα που ετέθηκαν ε, στα πλαίσια της νομοθετικής αυτής πρότασης και προσπάθησε επίσης με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο να έχει διάλογο για να λυθούν και τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει λόγω των διατάξεων της πρότασης αυτής με στόχο να ε, διασκεδάσει τις ανησυχίες που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο, τις νομικές συνέπειες και τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο ε, των ε, διατάξεων της νομοθετικής αυτής πρότασης, ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για τη στιγμή που ελπίζουμε ότι θα έρθει σύντομα, που το Συμβούλιο θα μπορέσει Ε, να ε, συγκεντρώσει την πολιτική βούληση όλων των μελών του, ώστε η νομοθετική πρόταση αυτή να υιοθετηθεί. Έχουμε εργαστεί ε, σε πολύ καλές συνθήκες με διάφορες προεδρίες. Με την Γαλλική και Σουηδική Προεδρία προσπαθήσαμε να Ε, ασχοληθούμε με κάποια από τα θεμελιώδη ζητήματα ε, της οδηγίας αυτής, ε, το πολύπλοκο θέμα του πεδίου εφαρμογής και των ορίων της ε, ευρωπαϊκής αρμοδιότητας. Μαζί με την Ισπανική και την Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου επικεντρωθήκαμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αναπηρία, την προσβασιμότητα και ε, την, τις λογικές προσαρμογές ε, που μπορούν να γίνουν για τέτοια άτομα, γνωρίζοντας ότι κάποια από τα κράτη-μέλη που ήταν κατά της πρότασης αυτής επικαλέστηκαν και το σημαντικό κόστος, το οικονομικό τις οικονομικές συνέπειες ε, για να συμμορφωθούν με την ε, πρόταση αυτή. Μαζί με την Βελγική Προεδρία εργαστήκαμε πάνω ε, στα στι χρηματοοικονομικές υπηρεσίε και την στέγαση. Με την ε, Πολωνική Προεδρία ε, σημειώσαμε πρόοδο όσον αφορά τι διακρίσει ε, λόγω ηλικίας, τα όρια ηλικία σε κάποιους τομείς. Μιλήσαμε για την εφαρμογή της οδηγίας σε ανήλικους και τη χρήση του, της ηλικίας ως παράγοντα κινδύνου στις ασφαλίσεις. Τον Μάρτιο του 2011 ε, είχαμε και ανάλογη ε, απόφαση του ΔΕΚ ε, στην υπόθεση Τέστασα και με την Δανέζικη Προεδρία ερευνάμε περαιτέρω το θέμα της ηλικία, το οποίο είναι ιδιαίτερα προβληματικό, ιδιαίτερα όσον αφορά την κοινωνική προστασία. Με χαρά μας είδαμε ότι όλες αυτές οι προεδρίες ε, κατάλαβαν την ανάγκη να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι, ώστε να παραμείνει ζωντανό το θέμα αυτό, αλλά με ουσιαστικό τρόπο, όχι μόνο με γραφειοκρατικό τρόπο. Προσπαθήσαμε να διασκεδάσουμε τις ε, παρανοήσεις και να διευκρινίσουμε τις διάφορες διατάξεις και τις συνέπειές τους για τη στιγμή που πολιτικά θα έχει οριμάσει ο χρόνος ώστε το Συμβούλιο να ε, ψηφίσει ομόφωνα την νομοθετική αυτή πρόταση. Επίσης, ε, συμμεριζόμαστε την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μόλις εξέφρασε ο εισηγητής και που έχει να κάνει με την ανάγκη να διατηρηθεί η ακαιρεότητα ε, της νομοθετικής αυτής πρότασης. Είναι μεγάλος ο πειρασμός να μειωθεί το πεδίο εφαρμογή της νομοθετικής αυτής πρότασης για να καλυφθούν οι ανησυχίες και για να βρεθεί ο ε, ελάχιστος ε, κοινός παρονομαστής. Αλλά έχουμε αντισταθεί στην, στον πειρασμό αυτόν έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε τους αρχικούς μας στόχους και να στοχεύσουμε σε ένα φιλόδοξο ε, μέσο το οποίο να εξυπηρετεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ε, ατόμων, των ανθρώπων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Κομισιόν αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή, την οποία ε, δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε. Η Κομισιόν θέλει να προωθηθεί ο φάκελος αυτός και να διατηρηθεί στην ακαιρεότητά του. Με το Συμβούλιο έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία. Ε, μερικοί θεωρούν ότι αυτά είναι απλά τεχνικά θέματα ε, και δεν θεωρούν ότι είναι σημαντικά πολιτικά θέματα. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι η πρόοδος σε τεχνικά ζητήματα είναι πολύ σημαντική. Κάποια επίμαχα σημεία παραμένουν και μπορεί να, χρειαστεί, να χρειαστεί πολιτική βούληση για να λυθούν, ε, αλλά χρειάζονται να γίνουν και απαραίτητες τεχνικές διευκρινήσεις. Επίσης είναι αλήθεια και το αναγνωρίζω αυτό, ότι η πρόοδος ε, σε τεχνικό επίπεδο δεν θα πείσει τα λίγα κράτη-μέλη που ε, έχουν θεμελιώδη αντίθεση απέναντι στην νομοθετική αυτή πρόταση για πολιτικούς λόγους. Τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο αυτό. Και πάλι, δεδομένη στις ανάγκη για ομοφωνία στο Συμβούλιο, χρειαζόμαστε μια πρακτική προσέγγιση και σοφή προσέγγιση. Η δουλειά μας πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόοδο σε τεχνικό επίπεδο ε, εφόσον ε, δεν ε, βλέπουμε στον ορίζοντα πολιτική ομοφωνία. Αλλά ε, μια συζήτηση όπως αυτή που ε, έχει οργανώσει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντική. Τέτοιες συζητήσεις θα είναι σημαντικές και στο εγγύς μέλλον. Και η πίεση από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τις κυβερνήσεις τους ε, για την προώθηση αυτού του νομοθετικού θέματος είναι πολύ σημαντική. Σημαντικό είναι και οι ενδιαφερόμενες ομάδες ε, να πιέζουν όχι μόνο το Συμβούλιο ως θεσμικό όργανο, αλλά και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Ε, η ήπια πίεση και διάλογος ε, με τις αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη είναι επίσης πολύ σημαντικά. Ο χρόνος ε, περνάει, αυτό είναι κοινότοπο, αλλά αυτό έχει αρνητικές ε, συνέπειες. Μερικές φορές όμως επιφέρει ε, τροποποιήσεις στις τοποθετήσεις διαφόρων κυβερνήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η θέση των ομάδων ενδιαφερομένων είναι πολύ σημαντικά για να διατηρηθεί η πίεση αυτή. Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη διατήρηση, θα συμβάλλει στη διατήρηση της, πίεσης, της πίεσης και ε, μόλις ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρία σε πολιτικό επίπεδο η Κομισιόν θα είναι έτοιμη ε, για να ε, εγκριθεί η πρόταση. Σε μια τέτοια στιγμή θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να έχουμε ολοκληρώσει το θέμα του αυτού. Κύριε Πρόεδρε, να κλείσω λέγοντας ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξή της προς οποιαδήποτε Προεδρία κεντρώνοντα σε θέματα ε, σημαντικά πάνω στα οποία θα πρέπει να εργαστούμε. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Ντορντέα. ακούσουμε τώρα την κυρία Άνε Μέτε και Αρχέ που εκπροσωπεί τη Δανέζικη Προεδρία. Δέκα λεπτά αν είναι δυνατόν, ώστε να έχουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Λόπες Αλγκυλάρου, τον εισηγητή για την οδηγία περί καταπολέμησης των διαδικασιών, τον κύριο Ρωμέβα. Ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα στην Επιτροπή ΛΥΠ. Χαίρομαι που ακούω πόση σημασία έχει για σας η πρόταση. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για τα στις αρχικέ παρατηρήσει, ε, δεν είμαι ότι θα κατορθώσω να μιλήσω ε, για 10 λεπτά και έτσι θα έχετε περισσότερο χρόνο για να θέσετε ερωτήσεις. Ε, δεν είναι και τόσο κακό αυτό. Παρακολουθώ το θέμα από την αρχή από το 2008 όταν η Κομισιόν κατέθεσε την πρότασή της, την παρακολούθησε κατά των προεδριών που ακολούθησαν και όπως γνωρίζετε μεγάλος αριθμός ανυψοποιών ε, ε δέχθηκαν ε, ευμενώς αυτή την πρόταση. Εγώ προσωπικά και η χώρα μου υποδέχθηκε ευνοϊκά την οδηγία αυτή περί της καταπολύμησης των διακρίσεων Από το 2008 λοιπόν ε, οι περισσότερες αντιπροσωπείες ε, δήλωσαν ε, την ανάγκη για ίση μεταχείριση ως μία από τις βασικές θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιπροσωπείς επίσης δήλωσαν την σημασία που έχει η σύνδεση αυτής της οδηγίας με την ε, με την ε, οδηγία του ΟΗΕ για το θέμα ε, της αναπηρίας και επίσης υπήρξαν κάποιες ελισσοπίες που έχουν επιφυλάξεις γενικής φύσης, κάτι που τόνισε και ο εισηγητής και η Κομισιόν, κατά πόσον αυτή η οδηγία θα μπορούσε να επηρεάσει τις, και να είναι αντίθετη προς τις εθνικές νομοθεσίες ε, κάποιες άλλες ερωτησίες ε, εξέφρασαν ανησυχίες αναφορικά με την έλλειψη ασφάλειας δικαίου σχετικά με τις εθνικές ε, συνέπειες της εν λόγω πρότασης ε, σε ό,τι φορά τώρα την Δανική Προεδρία. Κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας αφορήσαμε να συνεργαστούμε με την Πολωνική Προεδρία για το θέμα των διακρίσεων λόγω ηλικία. Στάλει τότε ένα ερωτηματολόγιο στα κρατημέλη, μέσω του οποίου ρωτούσαν κατά πόσον ε, θα μπορεί να υπάρξει πρόεδρος στο ζήτημα αυτών των ε, διακρίσεων λόγω ηλικία. Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε λοιπόν τι γραμμέ που είχε χαράξει η Πολωνική Προεδρία, διότι θεωρούμε ότι η πρόταση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θέλουμε να πετύχουμε πρόοδο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, ε, αλλά είμαστε και ρεαλιστές ε, παράλληλα. Φοβάσισαμε ως εκ τούτου να ακολουθήσουμε τα βήματα της Πολωνικής Προεδρίας και να ε, εργαστούμε πάνω στο ζήτημα της ηλικία όπως είπε ο κ. Δοντέα. Εδώ βρισκόμαστε προς το παρόν και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Παρατήρησα πως ο εισηγητής κ. Ρωμέβα έθεσε δύο ερωτήσει προς το Συμβούλιο. Μία από αυτέ ήταν η έλλειψη διαφάνειας. και ότι οι συνεδριάσεις είναι κλειστές, κάποια κράτη-μέλη είναι υπέρ, κάποια κατά, αλλά δεν δηλώνουμε ποια είναι κατά, ποια είναι υπέρ. Η στάση μου είναι αρκετά ένεκτη και η θέση μου λοιπόν είναι ανοιχτή. Βλέπω ότι κάθε εξάμεινο ε, υπάρχουν κάποιες δημοσιοποιήσεις. Υπάρχει λοιπόν επιθυμία ανοίγματο ε, για την σχετική οδηγία και η Ιδανική Προεδρία ε, η στάση που κρατάμε μέχρι σήμερα είναι να είτε κρατάει τα πράγματα όσο πιο διάφανα γίνεται και πώς ε, τώρα μπορεί το Κοινοβούλιο να βοηθήσει για την απεμπλοκή αυτής της πρότασης. Ωραία ερώτηση, αλλά και περίπλοκη συνάμα, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Ένας τρόπος είναι να πιέσουν προς την κατεύθυνση αυτή και να μας βοηθήσετε για την εξέβρεση κάποιων λύσεων. Νομίζω ότι αυτά εγώ να πω ως αρχικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ εκ νέου που με προσκαλέσατε στην συνεδρίασή σας, Πρόεδρος. Ευχαριστώ που ήσασταν σύντομοι. Και τώρα έχουμε τον γύρο των ερωταποκρίσεων. Κάποια, κάποια εκδηλώθηκαν ήδη, κύριε Χέτσον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι προφανές Συγγνώμη αν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι αυτές οι διαφορές που υπάρχουν οφείλονται στην Ευρώπη σε κάποια κινήματα της άκρας δεξιάς και όχι μόνο. Ε, το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό το οποίο συνέβη στις κάτω χώρες. με την ιστοσελίδα του Φιλελεύθερου Κόμματος ε, το οποίο παροτρύνει στην ε, ρατσιστική βία. Και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Απλά αυτό είναι το πλέον πρόσφατο. Είδαμε και περιπτώσεις ε, ξενοφοβίας, ε, διακρίσεων και θεωρώ ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις έχουν κάτι το κοινό. Και ότι οι αντιδράσεις ε, των κυβερνήσεων δεν είναι οι κατάλληλες, είναι αδύναμες. Ε, να σας αναφέρω και ένα άλλο παράδειγμα πάλι για την Ολλανδική κυβέρνηση που δεν ε, αντέδρασε καταδικάζοντας τα όσα δηλώνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεδομένου ότι το κόμμα αυτό συμμετέχει στον κυβερνητικό στασισμό. για ερώτηση μου εξή. Πιστεύετε ότι οι συνέπειε τη μελλοντική οδηγία σχετικά με το πώς οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διαχειριστούν το ζήτημα της παραβίασης θεμελιώδη δικαιωμάτων θα είναι θετικά η ανταπόκριση. Πιστεύετε με άλλα λόγια ότι η οδηγία αυτή θα μας βοηθήσει στο να μπορέσουν να αντιδράσουν κατάλληλα οι κυβερνήσεις και μια δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Τσουπάν Ντόρντα. Είσαστε εξοικειωμένος με το θέμα της Ένταξη των Ρώμα στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών, διότι θέλουμε, με άλλο γνωρίζουμε ότι αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω από τις εθνικές κυβερνήσεις. Πότε πιστεύετε λοιπόν ότι η Κομισιόν θα είναι σε θέση να υποβάλει μια συνολική έκθεση που θα αφορά στις απαντήσεις των εθνικών κυβερνήσεων για το θέμα των Ρώμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Εντσίου. Ο κύριος Κλέης. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής μα μίλησε για διαφάνεια. Ε, Είπαν ότι με νύχια και με δόντια Μερικέ χώρε ήταν κατά τις οδηγίες και προσπαθούν να την ε, τορπιλήσουν. Δεν ξέρω όμω ποια είναι αυτά τα κράτη-μέλη. Η εκπρόσωπος της Ιταλικής Προεδρίας επίσης μας μίλησε για διαφάνεια. Λοιπόν, αν είστε κι εσείς υπέρ της διαφάνειας, κατανομάστε αυτά τα κράτη που μπλοκάρουν την οδηγία. Για να διαμορφώσουμε και μια σαφέστερη εικόνα για το τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Ποια είναι τα κράτη-μέλη που είναι κατά της οδηγίας, κατά της εφαρμογής αυτής της οδηγίας και τι επιχειρήματα επικαλούνται αυτά τα κράτη-μέλη για να αντιταχθούν στην οδηγία. Εύκολα να τα συζητούμε αυτά, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι κάπως μονομερής αυτή η συζήτηση. Η οδηγία αυτή κανονικά θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη, αν εγκριθεί. Αλλά όλα αυτά γίνονται πολύ θεωρητικά. Η συζήτηση αποκτά ένα γενικό και αφηρημένο χαρακτήρα, γιατί δεν ξέρουμε καν ποια είναι τα κράτη-μέλη που είναι κατά της οδηγίας. Επίσης φαίνεται να δημιουργείται μια σύγχυση μεταξύ της οδηγίας κατά των διακρίσεων και της προσπάθειας ορισμένων χωρών να ελέγξουν τις μεταναστευτικές ροές. Φυσικά έχουμε την ιστοσελίδα του ΠΒΒ, του Κόμματος Ελευθερίας, στις ε, κάτω χώρες που ε, εξυμνεί το, τη μισαλοδοξία και το συζητήσαμε αυτό στις κάτω χώρες, αλλά το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί η οδηγία. Μας ενδιαφέρει μια συζήτηση που δεν θα είναι γενική και αόριστη. Ελπίζω μετά το πέρας της ακρόας αυτής να διαμορφώσουμε μια καλύτερη εικόνα, να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να εντοπίσουμε τις αντιφάσεις αυτής της νομοθεσίας με άλλα δικαιώματα που κατοχυρώνονται, όπως είναι της ελεύθερης έκφρασης. Ή αν μιλούμε για περιοριστική μετα... μεταναστευτική πολιτική, δεν θα πρέπει με το που επικαλούμαστε κάποιους περιορισμούς στη μετανάστευση αμέσως να μας κατηγορούν για υπέρμαχους των διακρίσεων. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι και ο κύριος Ρωμέβα θέλει να υποβάλει ερωτήσεις σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Πολύ σύντομα όμως. Η ερώτησή μου προς το Συμβούλιο είναι εξή. Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οι περισσότερες, αν όχι όλες οι τεχνικές και νομικές ε, επιφυλάξεις, οι ανησυχίες των κρατών μελών έχουν αποσοβηθεί και διευθετηθεί. γιατί είδαμε και τι πιθανές αντιφάσεις ε, θα δημιουργηθούν μεταξύ αυτής της ε, νομοθεσίας και των εθνικών διατάξεων και της εφαρμογής της. Από τη στιγμή που τα τεχνικά προβλήματα έχουν επιληθεί, ποια είναι τα επιχειρήματα που εξακολουθούν να επικαλούνται τα κράτη-μέλη για να μπλοκάρουν περαιτέρω την οδηγία, αν δεν υπάρχουν πια ούτε νομικά ούτε τεχνικά κολλήματα. Ποιος από τους προσκεκλημένους μας θέλει το λόγο γιατί κάποιες ερωτήσεις ε, απο... απευθύνθηκαν στο Συμβούλιο, άλλες στην Επιτροπή. Η κυρία Χέσελάγκερ, σε ό,τι αφορά την ερώτηση το κατά πόσο αν εγκριθεί η οδηγία αυτή θα, έχει, θα τον τρόπο τον οποίο οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν το θέμα της διάκρισης. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή είναι αναφυσβήτητα σοβαρή και πολύ σπουδαία και γι' αυτό είναι και τόσο χρονοβόρη διαδικασία, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντική η πρόταση και θα έχει επιπτώσεις ε, στην εθνική νομοθεσία. Θα έχει τεράστιο αντίκτυπο αν τελικά εγκριθεί. Και φυσικά εφόσον θα την εφαρμόσουμε κιόλα. Ο κύριος Κλέης εξέφρασε κάποιο προβληματισμό για τη διαφάνεια. Εγώ είπα ότι είμαστε αρκετά διαφανείς, δεν είπα ότι είμαστε τελείως διαφανείς. Κάποια κράτη, δεν είναι καθόλου μυστικό, αντιστέκονται στην πρόταση αυτή, ε, επικαλούμενοι την αρχή της επικουρικότητας και την αναλογικότητα, αλλά και τις νομικές και οικονομικές επιπτώσεις της πρότασης αυτής, της εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Σε ό,τι φορά τα σχόλια του εισηγητή του κ. Ρωμέβα, δεν νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στην πρόταση. Ε, σε ό,τι φορά την άρση των τεχνικών κολλημάτων. Υπήρξαν ε, κάποια προβλήματα που επιλύθηκαν από το 2008, αλλά εκκρεμούν και κάποια άλλα τεχνικά ε, θέματα. Δεν είναι ότι έχουν αρθεί όλα τα τεχνικά κολλήματα και απομένουν μόνο τα πολιτικά. Υπάρχουν ακόμη κάποιες τεχνικές εκκρεμότητες. Επίσης, είπα, ακούσαμε ότι ε, επί Ισπανικής ε, Προεδρίας ήταν πολύ πιο έντονη η ορμή και το δυναμικό που είχε δημιουργηθεί. Στο μεταξύ έχει κολλήσει κάπως η πρόταση, τα κράτη-μέλη είναι πιο απρόθυμα. Έχω την αίσθηση ότι όταν ε, εξετάζουμε αυτή την πρόταση, τα κράτη-μέλη έχουν ε, προβλήματα ως προς το εύρος, την εμβέλεια των τεχνικών επιπτώσεων και ως προς το βάθος των ε, διαφόρων προτάσεων. Εκεί λοιπόν θα πρέπει ε, να γίνει ακόμη κάποια επεξεργασία και να δούμε ποιες θα είναι οι πολιτικές επιπτώσεις, αν ο μόνος λόγος των επιφυλάξεων είναι οι πολιτικές επιπτώσεις. Δεν ξέρω αν σας φώτισα, σας διαφώτισα αυτά από το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ, συμφωνώ και εγώ με την Προεδρία, ότι δηλαδή αυτή η νομοθετική πρόταση θα έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις εφόσον υιοθετηθεί για την καθημερινότητα των πολιτών και για τη ζωή των πολιτών, γιατί θα έχει συγκεκριμένα ωφέλη για αυτούς και θα εξασφαλίσει καλύτερη νομική προστασία. Σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει του κυρίου Έντσιου, θα ήθελα να πω εν συντομία ότι κάποια από τα θέματα που έθιξε όντως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή της συγκεκριμένη οδηγίας. Αλλά κάποια άλλα θέματα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης πλαισίου του 2007 για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Πρόκειται βέβαια για μια απόφαση που προηγείται τη συνθήκη Λισαβόνα και με βάση τι διατάξει τη συνθήκη Λισαβόνα, μέσα σε μια πενταετία από τη θέση ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα, οι αποφάσει πλαίσιο που δεν έχουν λισαβονοποιηθεί εντό εισαγωγικών, όπω λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτομάτω ε, θα ε, εξομοιωθούν με οδηγίες. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει αμέσω να ξεκινήσει διαδικασίε επί παραβάση με βάση αυτές τις αποφάσεις πλαίσιο. Νομίζω ότι τα ερωτήματα του κυρίου Κλάης απαντήθηκαν. Τα πιο συχνά επιχειρήματα των κρατών μελών που αντιστέκονται στην πρόταση αφορούν την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Οπότε θα πρέπει να προταχθούν εδώ και πολιτικά επιχειρήματα υπέρ της οδηγίας και να ε, διεξαχθεί και ένας πολιτικός διάλογος. Συμφωνώ πάντως με την Προεδρία, με τη Δανική Προεδρία, ότι ναι με κάποια τεχνικά κολλήματα έχουν αρθεί, αλλά υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες και θα πρέπει να διευκρινιστούν άλλα τεχνικά θέματα δεν είναι μόνο πολιτικές ε, οι εκκρεμότητες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επεξεργαστεί και τα δύο στοιχεία, και το τεχνικό και το πολιτικό. Ε, ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Δεν βλέπω ε, να υπάρχει κανείς άλλος που να ζητάει τον λόγο. Να προχωρήσουμε λοιπόν στην πρώτη ουσιαστική συζήτηση στο πρώτο πάνελ μας που έχει να κάνει με το παρόν πεδίο εφαρμογή και του περιορισμούς ε, της ε, ισότητας ε, και του νόμου κατά των διακρίσεων. Έχουμε τον χάρτη δικαιωμάτων της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και την σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σήμερα λοιπόν τώρα εδώ θα εξετάσουμε Ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο για να αξιολογήσουμε το πεδίο εφαρμογή και τους περιορισμούς που υπάρχουν και θα επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 19 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρεις ε, ομιλητές έχουμε, διότι ενημερωθήκαμε ότι ο κύριος Ολιβιέντε Σούτερ από το Πανεπιστήμιο της Λουβέντε θα μπορέσει να είναι παρόν σήμερα. Έχουμε λοιπόν τρεις ομιλητές. Τον κύριο Ιωάννη Δημητρακόπουλο. Ζητά συγγνώμη ο πρόεδρος που δεν πρόφερε σωστά το όνομα. Παρακαλώ. από την Υπηρεσία Θεμελιωτών Δικαιωμάτων, ε, είναι επικεφαλής του Τμήματος για την Ισότητα και τα Δικαιώματα των Πολιτών. Την κυρία Ιζαμπέλ Σοπέν, που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, Νομικών Επιρογνωμόνων στον τομέα της, των μη διακρίσεων και τον κύριο Πιέρ Μποσσόν, Διευθυντή της Κοινωνικής Πλατφόρμας. Τρεις ομιλητές έχουμε. για το επόμενο δύο ώρο σχεδόν μέχρι τις 10 και 40 θα ακούσουμε τους ομιλητές μας από τις 10 και 40 μέχρι τις 11 και 10. Θα έχουμε έναν δεύτερο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Ξεκινάμε λοιπόν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 που καλέσατε τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, να συμμετάσχει στις ε, συζητήσεις σας για το πώς, μπορεί να πώς μπορούν να βελτιωθούν τα ε, νομικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθηθεί σε μεταχείριση και να παρασχεθεί αποτελεσματική προστασία κατά των διακρίσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι οδηγίες δεν δίνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για όλους τους λόγους διακρίσεων ε, οι διακρίσεις ε, λόγω θρησκείας, ε, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετικών προτιμήσεων είναι, για τους λόγους αυτούς υπάρχει προστασία μόνο στον τομέα της απασχόλησης. Ε, θέλουμε να, ε, δίνετε, να παρέχετε προστασία αντίστοιχη με ε, αυτήν που παρέχεται στην προστασία στην οδηγία για την φυλετική ισότητα. Στην παρουσίασή μου σύντομα θα σας δώσω κάποια παραδείγματα που έχουν να κάνουν με τις ε, με τον γενετήσιο προσανατολισμό, την, ε, τις αναπηρίες ε, και την ηλικία. Το 2009 ο οργανισμός κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσίασε την έκθεσή του σχετικά με τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ε, ε, φυλετικής ταυτότητας. Ε, βλέπουμε ότι γίνεται παρενόχληση όχι μόνο στον χώρο εργασία, αλλά και στα σχολεία και σε οίκους ευγυρίας όταν ζητά κανείς περίθαλψη για τον ίδιο ή για τον εταίρο του. Στην Δανία μια μελέτη του 2009 διαπίστωσε ότι το 16% των ατόμων ΛΟΑΔΗ είχαν ε, αυτοκτονήσει και 11% είχαν ε, προσπαθήσει, το οποίο είναι το διπλάσιο από τον ε, γενικό πληθυσμό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2008 μια μελέτη έδειξε ότι οι μισοί ομοφυλόφιλοι καλύπτουν, κρύβουν τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Επίσης, σε έκθεση του 2009, το 90% ε, των ε, ε, μαθητών που παρενόχλησαν στο σχολείο. Η παρενόχληση αυτή γίνεται επειδή είτε είναι είτε επειδή θεωρείται ότι τα παιδιά αυτά είναι ομοφιλόφιλα. Στη Φιλανδία σε έκθεση του 2011 για μειονότητες και τις διακρίσεις στην εκπαίδευση. Το 36% ε, των ε, αυτών που απάντησαν ε, είπαν ότι κάποια στιγμή είχαν υποστεί εκφοβισμό στα σχολεία λόγω του γενετήσου προσανατολισμού τους. Το να γίνονται αόρατοι οι άνθρωποι αυτοί γίνεται μια στρατηγική για να επιβίωσης και αυτό οδηγεί και σε χαμηλό αριθμό των παραπώνων για διακρίσεις λόγω γενετήσου προσανατολισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με, τα, τις προσφυγές για διακρίσεις για άλλους λόγους. Ένας αριθμός κρατών μελών, ε, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη προστασία, ήδη έχει βελτιώσει ε, την ε, νομοθεσία τους για την ίση μεταχείριση. Σε 18 κράτη-μέλη έχει επεκταθεί η νομοθεσία ώστε να καλύπτει και, την, και το γενετήσιο προσανατολισμό. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα ακαδημαϊκό δίκτυο ε, εμπειρογνωμόνων για τις αναπηρίες, ΑΝΕΔ, που έχουν συλλέξει ε, σημαντικό όγκο στοιχείων που δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για προστασία λόγω διακρίσεων, η προστασία κατά των διακρίσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, σε έκθεση για την εκπαίδευση των ε, ατόμων με αναπηρίες ε, στην Ευρώπη διαπιστώθηκε ότι ε, τα άτομα αυτά έχουν χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με τους μη αναπήρου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο το 15% των σπουδαστών με αναπηρίε, λαμβάνουν 5 ή περισσότερα GCE σε σχέση με το 80% αυτών που δεν έχουν αναπηρίε. Στην Αυστρία, οι φοιτητέ με αναπηρίε εγκαταλείπουν τις σπουδές μετα την 8 η ταξη αλλαζουν πηγαινουν σε ειδικο σχολειο επισης οι σπουδαστέ με αναπηριες μπορουν επισης να εγκαταλειπουν την δευτεροβαθμια εκπαιδευση προτου να μπορεσουν να φτασουν στο σημειο που επιτρεπεται η είσοδό τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ε, η έκθεση του Βούλγαρου ε, διαμεσολαβητή του 2010, του συνηγόρου του πολίτη, ε, έδειξε ότι υπήρχε έλλειψη προσβασιμότητας και σε νοσοκομεία, σε τμήματα κοινωνικής βοήθειας, σε οίκους ατόμων με αναπηρίες, καθώς και στις δημόσιες μεταφορές. Το 2010 το Ανώτατο Δικαστήριο της Βουλαρίας επιβεβαίωσε μια απόφαση ότι το Υπουργείο Υπουργείο Παιδείας ε, είχε ε, κάνει διακρίσεις ε, λόγω αναπηρίας επειδή δεν είχε διασφαλίσει την προσβασιμότητα παιδιών με ειδικέ ανάγκες. Και πρόσφατα το Ρουμανικό Εθνικό Συμβούλιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων ξεκίνησε νομική διαδικασία κατά ενός nightclub που αρνήθηκε την πρόσβαση σε γυναίκα που ήταν σε αναπηρικό καρεκλάκι. Κατά τη διάρκεια του 2011, μια σειρά κρατών μελών εισήγαγαν ε, τροποποίηση στην ομοθεσία και νέε πολιτικέ πρωτοβουλίε ε, έγιναν ε, για να αντιμετωπιστεί οι διακρίσει λόγω αναπηρία. Πολλά από αυτά ήταν αποτέλεσμα των προσπαθειών που έχουν γίνει να εφαρμοστεί πλήρω η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση. Για παράδειγμα, η Ισπανία υιοθέτησε νέα νομοθεσία τον Αύγουστο του 2011, ώστε η εθνική νομοθεσία να ευθυγραμμίζεται με τις ε, απαιτήσει ε, του CRPD των Ηνωμένων Εθνών που ε, συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, την κοινωνία των πολιτών και την κοινωνική προστασία. Η Σλοβενία στο τέλο του 2010 υιοθέτησε νομοθεσία που θεσπίζει την απαγόρευση διακρίσεων λόγω αναπηρίας από δημόσιε αρχέ όταν ασκούν τι αρμοδιότητε του. Αυτή η νομοθεσία απαγορεύει διακρίσεις σε πρόσβαση σε ε, αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα προς το κοινό. Και ε, θεσπίζει επίσης ε, την εξάλληψη εμποδίων που παρεμποδίζουν την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Το Σουηδικό Υπουργείο Ισότητας εξέδωσε μνημόνιο του τον Ιούλιο του 2012 που επεκτείνει την απαγόρευση διακρίσεων εις βάρος ανθρώπων με ε, αναπηρίες σε όλους τους τομείς πέρα από την ε, απασχόληση. Δηλαδή μιλάμε για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, σε, ε, ε, υγεία, περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες. Επίσης η ηλικία αποτελεί σημαντικό λόγο διακρίσεων στην έκθεση του 2011 ο ε, οργανισμός ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός ε, Υγείας λέει ότι οι διακρίσεις λόγω ηλικίας γίνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πρόσφατη ανάλυση δείχνει ότι οι διακρίσεις λόγω γύρανση ε, είναι οι πιο ε, συνηθίσεις στην Ευρώπη. Το 64% όσων απάντησαν ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με 44% σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι οι διακρίσεις λόγω γύρανσης είναι πολύ σημαντικές. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να αναφερθώ ε, σε μια σημαντική διάσταση των διακρίσεων, ή πολλαπλές διακρίσεις. Παρά την ε, αναγνώριση του κοινωνικού αντικτύπου λόγω, ε, της λόγω των πολλαπλών διακρίσεων, ο νόμος έχει αργήσει να ανταποκριθεί στο θέμα αυτό. Οι διακρίσεις για πάνω από ένα λόγους δείχνουν ότι ε, οι λίγε περιπτώσει όπου ε, αντιμετωπίζονται αυτές τι περιπτώσεις ε, δείχνουν ότι ο νόμος έχει μείνει πίσω στον τομέα αυτών. Πρόσφατες έρευνες του οργανισμού μας έχουν ε, ε, δώσει ε, επιπλέον στοιχεία για την ευάλωτη θέση, για παράδειγμα, των γυναικών μεταναστών στην πρόσβαση στην περίθαλψη. Γι' αυτό σημαντικό είναι κατά διάρκεια των συζητήσεών σας να λάβετε υπόψη τη δυνατότητα για αποτελεσματική νομική προστασία κατά των πολλαπλών διακρίσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ακριβώς την ώρα σας. Η κυρία Σοπέν έχει το λόγο για 10 λεπτά που θα μας παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμών σε θέματα διακρίσεων. Μου ζήτησαν να κάνω μια παρουσία σχετικά με τη μεταφορά των ε, δύο οδηγιών κατά των διακρίσεων. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφερόμενοι σε ε, ένα, κάποια αισιόδοξα μηνύματα. Στην αρχή υπήρχε μια πρωτοβουλία standing light, δηλαδή μετά την υιοθέτηση της οδηγίας ε, για κατά διακρίσεων ήταν ε, μια οργάνωση κοινωνίας των πολιτών, την οποία υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με εξαιρετική συνεργασία με την Κομισιόν. Το αναφέρω αυτό, διότι εδώ είμαστε ε, οι οργανώσεις, ε, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και ομού εγκρίναμε την οδηγία κατά των διακρίσεων. Να σας πω ότι στις αρχές του 90 όταν αρχίσαμε να συζητάμε, κανείς ποτέ δεν θα πίστευε ότι θα το πετυχαίναμε. Τώρα, όπως ο κύριος ε, Τσομπάν είπε, ε, οι πιέσεις δεν πρέπει να γίνουν μόνο προς το Συμβούλιο, αλλά χρειάζεται να γίνουν και στις εθνικές κυβερνήσεις. Οι ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και οι βουλευτές θα πρέπει να εργαστούν επί τόπου με τις εθνικές κυβερνήσεις. Τώρα, με κάποια επισιοδοξία, να πω, να πω το εξή το ε, του 2000 υπήρχε ε, μια τάση ε, θετική, αλλά δεν μπορέσαμε να υποφέρθουμε από αυτήν τώρα. Οι οδηγίες που εγκρίθηκαν κατά των διακρίσεων και το πεδίο αυτό το οποίο είναι γνωστό, το 2000 ε, η Κομισιόν αποφάσισε να δημιουργήσει ένα δίκτυο και ο πρώτος ρόλος, ο ρόλος αυτής του δικτύου ήταν να παρακολουθήσει την εφαρμογή της οδηγίας και να χορηγεί ανεξάρτητες πληροφορίε βάσει τις οποίε η Κομισιόν θα αποφάσιζε κατά πόσο θα είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν διαδικασίες επί παραβάση. Οι ε, διαδικασίες αυτές που ξέρετε είναι διαδικασίες που κινούνται ε, κατά των χωρών μελών για μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας και μη εφαρμογή τη. Τα περισσότερα αυτά που θα σας πω στηρίζονται σε συγκριτική ανάλυση που κάνει το δίκτυο. Ε, δημοσιεύουμε πολλές εκθέσεις, θεματικές εκθέσεις και κάθε χρόνο γίνεται μια συγκριτική ανάλυση που αναλύει το βαθμό μεταφοράς των δύο οδηγιών κατά των διακρίσεων. Τώρα, πώς ε, μετέφεραν τις οδηγίες τα κράτη-μέλη. Χρησιμοποίησαν ποικίλε οδούς, ε, χρησιμοποίησαν τις τη μεταφορά ε, λέξη προς λέξη της ε, οδηγίας. Άλλες φορές ε, οι πράξεις αυτές καλύπτουν περισσότερα παιδιά από ότι η οδηγία και θα επανέλθω. Τώρα έγκριση ενός συνδυασμού δράσεων και πράξεων συγγνώμη και έγκριση τροπολογιών σε κάποια νομοθετήματα έγκριση συνδυασμού ε, ε, πράξεων ε, σε ζητήματα εργασιακά και μεταφορά της οδηγίας. Γενικά τα κράτη-μέλη εφάρμοσαν αστικό και εργατικό δίκαιο και υπάρχουν διάφορα κομμάτια νομοθεσίας όπως στην Λετωνία. Πολλά κράτη-μέλη αποφάσισαν μεταφέρουν την οδηγία αυτή σε, με, μία πράξη, κάτι το οποίο ήταν θετικό, διότι δεν κατακαιρματίζει την οδηγία. Τώρα έχουμε περάσει 10 χρόνια και τα κράτη τα οποία έχουν μακρά παράδοση σε δήματα ε, καταπολέμηση διακρίσεων όπως το Ενού Βασίλειο και οι κατοχώρες και έχουν διάφορες ε, νομοθεσίες σχετικέ. Τώρα εργάζονται για να ενοποιήσουν όλε όλες, όλες αυτές τις νομοθεσίες. Ε, το Ενού Βασίλειο το πέτυχε αυτό πέρυσι και οι κατοχώρες εργάζονται ακόμα για να συγχωνεύσουν τις ποικίλε νομοθεσίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ενοποίησή του σε μια ποιο είναι τα πεδία που καλύπτονται. Η οδηγία δεν ορίζει πεδία και πολλά κράτη αποφάσισαν να το εφαρμόσουν. Αποφάσιστηκε επίσης να μην περιορίσουν τον, την νομοθεσία. σε λόγους αλλά το περισσότερα κράτη-μέλη αυτό που επέλεξαν ήταν να διευρύνουν ε, τις ε, διατάξεις ε, και εκτός της εργασίας σε άλλα ζητήματα που προστατεύουν για θέματα, για θέματα θρησκείας, πεπιθήσεων, αναπηρίας κλπ, ηλικίας για άλλα. Έχουν πολλά κράτη με έναν ανοιχτό κατάλογο των οποίων συμπεριλαμβάνουν και άλλα χαρακτηριστικά όπως ε, γεννητής προσανατολισμός κλπ. Πρέπει λοιπόν να ζητάμε τους λόγους, διότι το, η οδηγία περί φιλετικής ισότητας ε, πάει πιο μακριά από το ζήτημα της εργασίας. Δεν ε, πρόκειται να ε, μιλήσω για θέματα που άπτονται φιλετικού θέματος, ε, αλλά ε, τα όρια μεταξύ της της φιλετικής διάκρισης, της διάκρισης λόγω πεπιθήσεων και θρησκείας είναι δύσκολο να διαχωριστεί. Ο αντισημιτισμός σε κάποια κράτη καλύπτεται από την οδηγία περί φυλετικής βίας σε άλλα κράτη καλύπτεται από την νομοθεσία περί θρησκείας. Και όπως είπε ο ε, εισηγητής υπάρχει διαφορετική ε, προστασία ανάλογα με τη χώρα στην οποία κατοικεί τώρα. Ε, πεποίθηση και θρησκεία δεν υπήρξε μέχρι τώρα κάποιος ε, ορισμός. Αυτό το οποίο βλέπουμε σε ό,τι αφορά διακρίσεις στα ζητήματα αυτά αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας ε, περί εργασιακής ισότητας ε, όπου υπάρχουν κάποιες απαιτήσει περί θρησκευτικών πεπιθήσεων να γίνονται αποδεκτές και θα δούμε ότι αυτό είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, ειδικά για άτομα τα οποία ανήκουν σε μια θρησκεία τα οποία θεωρεί ότι δεν, μπορεί, δεν γίνεται αποδεκτή η ομοφιλοφιλία. Το θέμα τώρα, τον, υπάρχει το θέμα των θρησκευτικών συμβόλων. κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα ε, αναφορικά με την εφαρμογή της οδηγίας. Τώρα για τις αναπηρίες ε, ακούσαμε και γνωρίζουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επικυρώσει την, ε, τη σύμβαση. Τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν προσδιορίζουν την αναπηρία και βλέπουμε ότι τι περισσότερες φορές ε, παίρνουν διαορισμοί από το ζήτημα της κοινωνικής ε, προστασίας και όχι από την ε, οδηγία για την κατάπολη των διακρίσεων. Ο κ. Τσεμπάν ανέφερε επίση το ζήτημα των τεχνικών προσαρμογών που αφορά στα άτομα με αναπηρίες. βλέπουμε ότι αυτές οι εύλογες προσαρμογές είναι δεκτές αλλά όχι με νομική πράξη. Παράδειγμα, εύλογες προσαρμογές που σχετίζονται με το θέμα των θρησκευτικών εορτών, αλλά μόνο δύο κράτη αποφάσισαν να τα συμπεριλάβουν στις νομοθεσίες. Το σεξουαλικό του αντολισμός ε, νομική προστασία για πρώτη φορά σε ό,τι φορά την γενετήσιο ε, προσανατολισμό. Με πολύ λίγα έχουν ε, ορίσει λόγω των δυσκολιών οι οποίες ε, οφείλονται στο εργασιακή νομοθεσία ηλικία θεωρείται ότι είναι ένα αντικειμενικό κριτήριο, αλλά αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, διότι τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν έχουν νομοθεσία για την καταπολύπτωση διακρίσεων λόγω ηλικίας. Υπάρχουν μια σειρά εξαιρέσεων και παραμένει σημαντική αβεβαιότητα αναφορικά με το τι μορφές διακρίσεων θα πρέπει να συμπεριληφθούν Νομίζω ότι υπάρχουν 15 αποφάσεις ε, του από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 9 ε, αποφάσεις ε, από τις 13 αφορούν από τις 13 αφορούν την διακρίση λόγω ηλικίας. Δεχόμαστε λοιπόν θετικά την αναφορά που γίνεται για τις πολλαπλές διακρίσεις. Οι διακρίσεις ε, μερικέ φορές ε, μπορούν ε, να αφορούν τα χαρακτηριστικά ενό προσώπου, τα οποία μπορεί να είναι μπορεί και να μην είναι σωστά. Η Κομισιόν θέλησε λοιπόν να καλύψει το θέμα των ισχυρισμών. Μόνο κάποια κράτη-μέλη αποκλείσανε στην νομοθεσία τους αυτές της διακρίσεις. Δεν θα πάω τώρα στο θέμα των το αντικειμένο ούτε το πεδίο. Θα σας αναφέρω ότι στον τομέα της εργασία υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές αναφορικά με θέματα της, ε, των ε, ελεύθερων απασχολούμενων, των απασχολούμενων. Σχετικά με την κοινωνική προστασία, πολλές διατάξεις υπάρχουν σε συγκεκριμένα νομοθετήματα που άπτονται των κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικής πρόνοιας εκπαίδευση περισσότερα κράτη-μέλη. Το ζήτημα αφορά περισσότερο στα παιδιά ε, ε, που ανήκουν σε μειονότητες ε, τις διακρίσεις που μπορούν να οφείλονται σε λόγους θρησκείας. Αυτό που δεν έχει ακόμα αποφασιστεί είναι εάν ε, εφαρμόζεται μόνο στους στο δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους. 24 κράτη από τα 27 έχουν εν, εντάξει τις ε, οδηγίες αυτές στο δίκαιό τους Σχετικά με τις ε, αποκλήσεις, τις εξαιρέσεις, ε, υπάρχουν πολλές ε, θετική δράση. Είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε τι είδους θετικές δράσεις προβλέπονται, αλλά τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει μέτρα θετικών δράσεων. Οι δύο τομείς είναι η αναπηρία και η εθνικότητα, η εθνότητα και η παιδεία. εφαρμογή των δύο οδηγιών έφτασε την στιγμή όπου τα κράτη -μέλη, ορισμένα κράτη-μέλη επέτρεψαν ε, τον ε, γάμους μεταξύ προσώπων δυο φιλου αλλά γεγονός είναι ότι σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν περιορισμοί για να λειτουργήσει πάνω λοιπόν αποτελεσματικά νομοθεσία χρειάζεται να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Καλό είναι να υπάρχει, υπάρχει νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται, δεν θα πρέπει να παραμένει νεκρογράμμα. δικαστικές και διοικητικές ε, διαδικασίες υπάρχουν σε περισσότερα κράτη-μέλη όπου περιλαμβάνεται και η διαμεσολάβηση και ο συμβασμός τα κράτη-μέλη έχουν διακριτική ευχέρεια για το πώς ε, θα υλοποιήσουν τις ε, οδηγίες ε, και υπάρχουν διαφορετικές, ε, διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής η δευτερεύουσα παράγωγη νομοθεσία μάλλον σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί να δημιουργηθούν κάποιοι φραγμοί όπως η λειτουργία των των υπηρεσιών για κάποια χρόνια προτού να μπορέσουν να ασκούν αποτελεσματικά το ρόλο τους κλπ. Ε, κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν ευθυγραμμιστεί ακόμα με τις οδηγίες. Ε, τώρα η θυματοποίηση είναι ε, σε ε, είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τον χρόνο εργασίας, αλλά τώρα και τα ένομα μέσα τα οποία υπάρχουν όπως οι αποζημιώσεις που μπορούν να χορηγηθούν σε περίπτωση διακρίσεων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να οδηγήσει μια διάκριση σε χιλιάδες ε, ε, λίρες αποζημίωση σε άλλα κράτη-μέλη είναι πολύ μικρότερη. Υπάρχουν, υπάρχει επίσης ε, και ελάχιστη νομολογία στα περισσότερα κράτη. Υπάρχουν κάποιοι φραγμοί για πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη. Ε, χρονικό, χρονικό διάστημα το οποίο ισχύει για τις καταγγελίες ε, οδηγεί σε κάποια προβλήματα, δημιουργεί εμπόδια πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Επόμενο σημείο είναι το σώμα ισότητας. Ε, αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε εδώ είναι ότι μόνο πέντε κράτη αποφάσισαν να περιορίσουν τις αρμοδιότητες ε, του φορέα ισότητας ε, τα, όλα τα υπόλοιπα, φορεί. φορείς έχουν διευρύνει τους, ε, το πεδίο δράσης σύμφωνα με την οδηγία για την εργασία. Χρειάζεται να αναφέρουμε ότι μόνο ότι δεν απαιτείται η ανεξαρτησία αυτών των φορέων, πρέπει όμως να αποδείξουν ότι λειτουργούν ανεξάρτητα. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η δράση τους περιορίζεται λόγω της οικονομικής κρίσης. Εμείς έχουμε στόχο να προωθήσουμε τις προφορίες, να προωθήσουμε την νομοθεσία κατά των διακρίσεων αλλά συχνά δεν έχουμε τα, ως φορείς τα απαραίτητα μέσα οικονομικά. Καταλήγοντας πω ότι πέραν του εργασίες υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία προστατεύονται οι πολίτες από τις αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Πάντως υπάρχουν κάποιες διαφορές, ε, κάποιες ελλείψεις. Θα έχετε το PowerPoint. Αυτό που θα πρέπει να προλάβουμε είναι οι πολίτες να μην προστατεύουν διαφορετικά στις κρατημένες. Αρχές του 1990, όταν ξεκινήσαμε, θεωρήσαμε ότι υπήρχαν προβλήματα στην ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και αυτό καλό Ευχαριστώ. Thank you so much. That's been a thorough explanation. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ εμπεριστατωμένη η παρουσίαση αυτή και πραγματικά κάνατε μια γενική επισκόπηση της κατάστασης και του δικαίου που ισχύει στα κράτη-μέλη από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Δικτύου ε, των Φορέων και των Νομικών Εμπειρογνωμών. Ο κύριος Πιέρ Μποσόν, που είναι διευθυντή τη κοινωνική πλατφόρμα. Η κοινωνική πλατφόρμα είναι το μεγαλύτερο δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τελευταία τέσσερα χρόνια δίνουμε μάχη για απεμπλοκή των εργασιών αυτή τη οδηγία. Υπάρχει αίσθηση του κατεπήγοντο, γιατί ο κόσμος περιμένει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά του, να μπορεί να σκίσει τα δικαιώματά του. Είναι κρίμα που έχει κολλήσει το θέμα στο Συμβούλιο. Και αυτό που ζητούμε πρώτα απ' όλα θα είναι η συνοχή. Αυτή, τη λέξη θα την ακούσετε πολλές φορές ε, στην ε, εισαγωγή μου, στην εισηγησή μου. Θέλουμε μία συνοχή στην αντιμετώπιση. Η συμπολίτε μα υποφέρουν από τι διακρίσει. Ένα στου έξι Ευρωπαίου υφίσταται διακρίσει. Σήμερα έχουμε γύρω στου 200 ε, στην αίθουσα. Αν σκεφτούμε ότι ένα στους έξι υφίσταται διακριτικές με, διακριτική μεταχείριση για να βάλουμε να καθίσουν όλοι μαζί, βλέπετε ε, πόσοι ε, εμπίπτουν σε αυτές τις διακρίσεις. Πάντως, πιστεύω ότι αν είχατε υποστεί διακρίσεις στο παρελθόν δεν θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε τις ε, καλές σπουδέ που κάνατε στο καλό πανεπιστήμιο και να βρείτε την καλή δουλειά. Ούτε θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση. Γιατί δεν θα είχατε καν ένα σπίτι να ζήσετε. Μία σκεπή πάνω από το κεφάλι σας γιατί οι τράπεζες θα αρνούνταν να σας χορηγήσουν ενυπόθηκο δάνειο. Επίσης, ε, ε, μπορεί ε, να, σας, να χτυπάει το BlackBerry κινητό σας γιατί σας τηλεφωνεί ο διευθυντής του σχολείου για να πει ότι το παιδί σας υφίσταται εκφοβισμό στο σχολείο από τους συμμαθητές του. Ένας άλλος λόγος διάκρισης θα είναι ότι έχετε βαρεθεί να συγκατοικείτε με τους φίλους σας, γιατί κάθε φορά που προσπαθείτε να νοικιάσετε για δικό σας λογαριασμό σας αρνούνται ε, το ενίκιο. Για όλους αυτούς τους λόγους ε, δεν θα μπορούσατε να είστε εδώ και βλέπετε πώς είναι οι λόγοι των διακρίσεων. Έχουμε κουραστεί πια, έχουμε απειδήσει να περιμένουμε τόσα χρόνια, τέσσερα χρόνια να εγκριθεί αυτή η οδηγία. Ο στόχος της νομοθεσίας ε, δεν είναι να αλλάξει την κατάσταση. Δεν πρόκειται να αποκατασταθεί μία ανοιχτή ισότητα, αλλά χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα νομικό πλαίσιο που να ε, κατοχυρώνει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται και σε περίπτωση διάκρισης να μπορεί κάποιο να διεκδικήσει αποκατάσταση. Γνωρίζουμε τι εστί κοινωνικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει. Πιστεύουμε στην ισότητα, έχουμε αξίε και αρχέ. Πιστεύουμε ότι όλοι είμαστε ίσοι και έχουμε ίσα δικαιώματα. Θα ήθελα τώρα να πάω προς την πλευρά του Συμβουλίου. Γιατί αυτό που μας ε, διαφέρει είναι η πολιτική βούληση που θα πρέπει να δείξει το κράτη-μέλη για να πετύχουμε την απεμπλοκή. Καταρχήν, πολιτική βούληση ποιου. Οι κοινωνικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει υποστηρίζουν την οδηγία. Το ίδιο και η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα συνδικάτα είναι υπέρ τη οδηγία στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι οι συμπολίτε μας, οι Ευρωπαίοι πολίτες, είναι υπέρ της οδηγίας αναφανδών. Ποιος λοιπόν είναι κατά της οδηγίας όταν μας λέτε ότι μερικά κράτη-μέλη είναι κατά της οδηγίας. Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να σα μεταφέρω είναι η συνοχή σε ό,τι αφορά του πολιτικού στόχου του Συμβουλίου. Το 2000, όταν η οδηγία για τι φυλετικέ διακρίσει εγκρίθηκε, μα είπαν ότι οφειλόταν ε, η έγκρισή τη στην κατάσταση στην Αυστρία. Εντάξει, το καταλάβαμε. Αλλά Είχαμε και άλλε προτεραιότητε όπω την απασχόληση στα πλαίσια τη στρατηγική Λισαβόνα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε απασχόληση για όλου. Θέλουμε ισότητα για την ισότητα, ε, ισότητα για την απασχόληση. Ε, από τη μια μα λέει θέλουμε ισότητα για την απασχόληση, από την άλλη δεν θέλουμε ισότητα για την ισότητα. Λίγη συνοχή λοιπόν παρακαλώ για πώς είναι δυνατόν ένα ε, νεαρό παιδί με αναπηρία που δεν πήγε σε σχολείο, γιατί δεν μπόρεσε να πάει σε κανονικό σχολείο, δεν μπορεί να ανεβεί στο λεωφορείο να πάει στη δουλειά του. Δεν μπορεί να μπει σε ένα τρένο να πάει στη δουλειά του. Πώ αυτό ο άνθρωπο θα, θα βρει δουλειά, Γιατί θέλετε ισότητα στην απασχόληση. Ε, να αποκαταστήσετε λοιπόν μια συνοχή. Με την οδηγία αυτή θα εξασφαλίσετε πρόσβαση των ανθρώπων στι υπηρεσίε. Χρειάζεται αυτή η πρόσβαση για να μπορέσει κάποιο να βρει δουλειά. Πέμπτο μήνυμα. Συνοχή με τη στρατηγική του Συμβουλίου που τάσεται υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Δεν συμφωνώ κατά ανάγκη με το στόχο αυτό. Θα είναι συζητήσιμο το θέμα. Θέλετε να μειώσετε την ανεργία, θέλετε να καταπολεμήσετε τη φτώχεια, θέλετε να εξασφαλίσετε απασχόληση. Αν βάλετε όμως ως πρωταρχικό στόχο σας την ισότητα, τότε ίσως καταφέρετε να υλοποιήσετε και τους υπόλοιπους στόχους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Γιατί γι' αυτό, αυτό μας ζητάει το Συμβούλιο, όχι μόνο αρχές και στόχους, αλλά και συγκεκριμένα παραδείγματα. Ανώτατη παιδεία στη Γαλλία. Όταν παίρνετε παιδιά από τα προάστια και μέσω ειδικών προγραμμάτων τα βάζετε στα πανεπιστήμια, ε, τα εξυπηρετείτε, γιατί δεν μένουν πια στα απροάστια που η φτώχεια είναι πολύ πιο έντονη, έχουν πρόσβαση στην, στα πανεπιστήμια, κάτι που δεν ισχύει προηγουμένω. και με ένα πτυχίο ανώτατη σχολή έχουν καλύτερη ε, πρόσβαση και στην απασχόληση. Αν λοιπόν έχετε την ισότητα στο πρωτοχικό στόχο, υλοποιείτε και του άλλου στόχου, όπω είναι η απασχόληση και η πρόσβαση η καταπολέμηση της φτώχειας. Ένα άλλο μήνυμα που είναι πολύ δύσκολο για μας να το αντιληφθούμε και είμαι ιδιαίτερα ενοχλημένο, είναι η συνοχή σε σχέση με άλλε νομοθετικέ διατάξει. Όταν μα λέει το Συμβούλιο ότι υπάρχουν προβλήματα αρμοδιότητα με την οδηγία, ότι υπάρχουν προβλήματα επικουρικότητα, παρακαλώ εξηγήστε μα πώ είναι δυνατόν το 2000 να εγκρίνεται την οδηγία για τις φιλετικές, κατά των φιλετικών διακρίσεων και ε, ενώ η συνθήκη τη Λισαβόνα το 2010 βελτιώνει και ενισχύει τις κοινοτικέ αρμοδιότητες, ξαφνικά λέτε ότι δεν υπάρχουν αρμοδιότητε, δεν υπάρχει κοινοτική αρμοδιότητα για να εγκρίνουμε αυτή την οδηγία. Εξηγήστε μα παρακαλώ, όπω. Σα ζήτησε και ο συγγητή ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα σήμερα το πρωί. Αναφέρθηκε και το θέμα του κόστους. Έχω μία ερώτηση. Μερικές φορές θα πρέπει να αξιολογούμε και να αποτιμούμε το κόστος της μη επένδυσης στην ισότητα και στην παιδεία. Από μία μελέτη στη Γαλλία φάνηκε ότι αν επενδύσουμε 1.000 ε, ευρώ σε κάθε φοιτητή, κάνουμε τεράστιες εξοικονομήσεις από επιδόματα ανεργίας, από άλλα κοινωνικά επιδόματα που θα χρειαστούν αν ο άνθρωπος αυτός δεν βρει δουλειά ή ε, ζει σε συνθήκες φτώχειας. Σε ό,τι αφορά τη συνοχή, θέλουμε συνοχή και με την δημοκρατική διαδικασία. Μερικέ οργανώσει, και εδώ όλε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, ε, λένε το ίδιο, μην αποφασίζετε για μας ερήμην μας. Συνεργαζόμαστε με το, συμβούλιο, με την, με το Κοινοβούλιο, με την, επι, με την Κομισιόν, με τα συνδικάτα. Έχουμε εκδώσει και κοινή δήλωση. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να συνομιλήσουμε και με εκπροσώπους του Συμβουλίου. Γιατί μας αποκλεί το Συμβούλιο, γιατί δεν μας αφήνει να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας με τους εμπειρογνώμονές μας. Θέλουμε να μάθουμε ποια τι προβλήματα έχει το Συμβούλιο για να μπορέσουμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις. Και θέλουμε και διαφάνεια, να δούμε πού ε, υπάρχουν προβλήματα, πού δημιουργούνται στενοποί. Τέλος, για ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό, έχουμε δυσκολίες και έχουμε επιβδίσει κιόλα. Θέλουμε η κοινωνία των πολιτών να αντιληφθεί ότι μία οδηγία κατά των διακρίσεων δεν πρόκειται να αποκαταστήσει την ισότητα, αλλά δημιουργεί κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε ένα πλαίσιο, κάποιες διατάξεις στην κοινωνία για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Και παρόλα αυτά φαίνεται ότι ακόμη και ένα τέτοιο πλαίσιο ελαχίστων είναι ε, Κάτι που δεν μπορεί να κάνει το Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε την οδηγία αυτή. Δεν πρόκειται να αλλάξει αν είναι μια ανοιχτή Ευρώπη χάρη σε αυτή την οδηγία. Αλλά ξεκινήστε τι διαπραγματεύσει σε πολιτικό επίπεδο και πείτε μα με σαφήνεια γιατί είστε κατά αυτή τη οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ποσό. Μπορούμε τώρα να έχουμε μια, ένα γύρο απαντήσεων. Πρώτα έχουν τη δυνατότητα τα μέλη της Επιτροπής μας να υποβάλουν ερωτήσεις στους πανελίστες. Θέλει κανείς το λόγο, παρακαλώ, η κυρία Λούνατσεκ, να σημειώσω τους ε, ομιλητές, γιατί αναφέρθηκαν ε, κάποια σχόλια για τις θέσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Φαντάζομαι ότι θα θέλουν να αντιδράσουν το Συμβουλίο και η Επιτροπή, αλλά πρώτα να ακούσουμε τις ερωτήσεις των μελών και του εισηγητού μας φυσικά. Κύριε Λούνατζεκ πρώτα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ε, εμπειρογνώμονές μας για τις ε, πολύ εμπεριστατωμένες και μεστές εισηγήσεις τους που ε, δείχνουν γιατί κάνουμε αυτή την οδηγία. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Έχουμε βαρεθεί να περιμένουμε. Χρόνια ολόκληρα έχει αποτελματωθεί η συζήτηση για την οδηγία αυτή. Θα πρέπει επιτέλους να δοθεί μια όθηση. Ο κύριος Μποσό μίλησε και για το κόστος. Μου άρεσε που είπατε να αποτιμήσουμε και το κόστος της μη εφαρμογής και όχι μόνο το κόστος της εφαρμογής, γιατί αυτό το παραβλέπουμε συστηματικά. Δεν παρακολούθησα το πρώτο τμήμα της δημόσιας ακρόασης. Δεν ξέρω λοιπόν αν αναφέρθηκε τελικά ποιες είναι οι χώρες που μπλοκάρουν την οδηγία. Αλλά ξέρω ότι μία από τις χώρες αυτές είναι η Γερμανία. Και είχα μία ε, ενδιαφέρουσα σύντομη συζήτηση ε, με τον κύριο Βέστεν Βέλε στις ε, Ευρωπαϊκές Αθλητικές Εκδηλώσεις Λεσβιών και Ομοφιλοφίλων. Είχε συνάντηση με τους συμμετέχοντες, ήμουν και εγώ εκεί. Και μάλιστα ρώτησα τότε γιατί η Γερμανία δεν θα εφαρμόσει την οδηγία αυτή, παρόλο που αν δεν κάνω λάθος ήταν και στη συμφωνία του συνασπισμού. Το ρώτησε λοιπόν γιατί ε, δεν προωθείτε αυτό το θέμα, γιατί και εσείς κύριε Βεστερβέλη είστε ε, δημόσια, έχετε δηλώσει είστε ομοφιλόφιλος. Και μου λέει ας αφήσουμε την πολιτική. Αυτά σας τα λέω ε, ανεκδοτολογικά. Πάντως στην ε, Γερμανία το επιχείρημα που προβάλλεται είναι το κόστος εφαρμογής όχι τόσο για τις διακρίσεις κατά, για το γενετι, λόγω γενετήσου προσανατολισμού, αλλά το, για τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Για να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές για καλύτερη πρόσβαση των αναπηρικών πολυθρόνων κτλ. Έχετε κάνει αποτίμηση όμως και του κόστου της μη εφαρμογής σε ορισμένες χώρες, γιατί νομίζω ότι αν δοθούν και αυτές οι αποτιμήσεις, ίσως... Ε, διασυστούν τα επιχειρήματα των κρατών μελών που επικαλούνται το κόστος. Γιατί αν ακούσουμε αυτή την κατάθλιψη, την, τη σκέψη αυτοκτονίας, ε, γενικώ την πολύ κακή ψυχική διάθεση και τα προβλήματα, την οδύνη που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που υφίστανται διακρίσεις. Κυρία Γκόντς. Άκουσα αυτούς από εσά που είπαν ότι χρειαζόμαστε αυτήν την οριζόντια οδηγία ε, κατά των διακρίσεων και ήταν πολύ ενδιαφέρον που ε, ακούσαμε τα σχετικά με την εφαρμογή, το πώς μεταφέρθηκε στην Εθνική Νομοθεσία των διαφόρων χωρών. Αλλά βλέπουμε όχι μόνο ελλείψεις κατά την εφαρμογή, ε, μερικές φορές έχω και την εντύπωση ότι οπισθοδρομούμε σε πολλές χώρες όσον αφορά την εφαρμογή. Ακόμα και όσον αφορά την οδηγία στον τομέα της απασχόλησης. Ε, και γι' αυτό κύριε Δημητρακόπουλε ήταν πολύ ενδιαφέρον που άκουσα από εσά ότι αυτοί που υφίστανται διακρίσεις δεν απευθύνονται στις αρχές, ακόμα και στις χώρες όπου υπάρχουν αυτοί οι φορείς ισότητας. Και νομίζω ότι αυτό συνδέεται στενά με το κοινωνικό κλίμα. με τους ε, πολιτικούς παράγοντες που δεν έχουν ε, εκφράσει την υποστήριξή τους ε, για την οδηγία αυτή κατά των διακρίσεων. Θα ήθελα να ακούσω λίγα περισσότερα από εσά σχετικά με το πώς βλέπετε την κατάσταση στην Ευρώπη. Αναφέρατε ότι το πολιτικό κλίμα ήταν πολύ σημαντικό κατά την υιοθεσία των οδηγιών αυτών. Εσείς πώς βλέπετε την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. No other hands are being raised. Να ακούσουμε από τον εισηγητή μας, ε, τον κύριο Ρωμέβα. Δύο ερωτήσεις έχω. Ε, ακούσαμε ξεκάθαρα κάποια στοιχεία υπάρχουν. Περισσότερα ακούσαμε μια σύνοψη ε, ήταν αρκετή, αρκετά πλήρης και αρκετά σαφής, αλλά δείχνει ακριβώς ε, την κορυφή του παγόβουνου. Η πραγματικότητα είναι ακόμα χειρότερη από αυτά που ακούσαμε. Έχουμε λοιπόν σαφή στοιχεία. Ακούσαμε επίσης τις δυνατότητες ε, και ε, την συμβασιμότητα με το, την εθνική νομοθεσία η πολιτική αντίθεση ε, στο να έχουμε εδώ ευρωπαϊκά πρότυπα ε, αντίκειται στο γεγονός ότι πολλά κράτη-μέλη ε, έχουν τα στοιχεία αυτά στην εθνική τους νομοθεσία. Γιατί λοιπόν να μην θέλουμε εθνική νομοθεσία. Θα ήθελα να ξέρω εάν αυτή η θέση μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση των ε, συνθήκων, ε, της νομολογίας του δικαστηρίου, του, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες. Υπάρχει χώρος Υπάρχει η ιδέα ότι ε, η αντίθεση στα ευρωπαϊκά πρότυπα μπορεί να παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Και τέλος, όσον αφορά αυτό που ανέφερε η Ουρρίκε. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να ομολογήσω ότι πολιτικά δεν νιώθω πολύ άνετα να χρησιμοποιώ το επιχείρημα του κόστους ε, σε ένα νομοθέτημα που έχει να κάνει με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα τέτοιο νομοθέτημα άσχετα από το κόστος. Αλλά επειδή εδώ και πολλά χρόνια ακούω αυτό το επιχείρημα, ε, το αντιεπιχείρημα είναι ας μιλήσουμε για το συνολικό κόστος ε, και γι' αυτό ζήτησα από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να μελετήσει το θέμα. Και ε, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, βαρεθήκαμε να ακούμε ε, το επιχείρημα ε, περί κόστους. Θέλουμε να γνωρίζουμε το κόστος, ναι, αλλά ας βάλουμε όλες τις δαπάνες στο ε, τραπέζι και να εξετάσουμε ποιο είναι το κόστος της μη εφαρμογής των διατάξεων αυτών. Τότε θα έχουμε σαφή εικόνα του του τι συζητάμε. Το να μιλάμε όμως μόνο για το κόστος των λογικών προσαρμογών ε, που πρέπει να γίνουν για άτομα με ειδικέ ανάγκες, με, με αναπηρίες, ε, νομίζω ότι είναι λάθος. Θα ήθελα ε, λοιπόν να συμφωνήσω με τη συνάδελφο Λουκατσέκ. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση στο θέμα. Ίσως η Κομισιόν και το Συμβούλιο θέλουν να απαντήσουν στις παρατηρήσεις που έγιναν από τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σε αυτά που ακούσαμε σχετικά με το μπλοκάρισμα της πρωτοβουλίας και την θέση κάποιων ε, κρατών μελών ή φορέων. Τότε να δώσω το λόγο στον κύριο Ποσάν πάλι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία σύντομη παρατήρηση σχετικά με το τι είπε η Ευρωβουλευτή ε, Λουκατσέκ για το κόστο. Δύο θέματα υπάρχουν εδώ. Ε, συμφωνώ με το θέμα του κόστου ε, των μη επενδύσεων. θα ήθελα όμω να επανέλθω στο θέμα τη επαφή ανάμεσα στο Συμβούλιο και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αναπηριών σε συζητήσεις που είχαμε μαζί συμφωνήσαμε ότι στο, στους ε, ε, διαδρόμους ακούσαμε ότι θα πρέπει ε, να να κατεδαφιστούν ολόκληρες κοινότητες και να ξαναχτιστούν για να είναι προσβάσιμες. Δεν μιλάμε όμως για κάτι τέτοιο. Δεν λέμε ότι η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχει, στο τραπέζι, να συμμετέχει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Έχουμε όμω κάποια εμπειρογνωμοσύνη, μπορούμε να υποβάλουμε κάποια έγγραφα, μπορούμε να συμμετάσχουμε σε δημόσιε ακροάσει όπω είναι η σημερινή, όπου μπορούμε να εξηγήσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για εφαρμογή τη οδηγία. Σα ευχαριστώ για την ελευθερολογία σα, η κυρία Σοπέν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο σχόλια. Το ένα το ανέφερε ο εισηγητής το κατά πόσο αντιβαίνει η οδηγία αυτή σε προηγούμενε οδηγίε. Θα πρέπει σίγουρα να γίνει και σχετική μελέτη. Αλλά από ό,τι φαίνεται αντιβαίνει και στη Σύμβαση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στη Σύμβαση του ΟΗΕ για την αναπηρία. Επανέρχομαι στη δεκαετία του 90, τότε που κάναμε εκστρατεία υπέρ της φιλετικής ισότητας και τη ε, θέσπιση νομοθεσία κατά των φυλετικών διακρίσεων. Και όταν αναφερθήκαμε στην αντιστροφή του βάρου απόδειξη, είχαν τρελαθεί όλοι και είπαν ότι είναι αδύνατο. Παρ' όλα αυτά το 1997 ε, ενέκρινε οδηγία που περιείχε και το, ε, την αντιστροφή του βάρους απόδειξης σε θέματα ισότητας φύλου. Κάτι δηλαδή που ίσχυε για την ισότητα των δύο φύλων δεν ίσχυε για τις φυλετικές διακρίσεις. Και Τώρα έχω την αίσθηση ότι αυτό που ισχύει για τις φυλετικές διακρίσεις δεν είναι αρκετά καλό, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις διακρίσεις λόγω αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσεω προσανατολισμού. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στα κράτη-μέλη τις υποχρεώσεις τους όταν εγκρίνουν, όταν κυρώνουν διεθνείς συμφωνίες ή συνθήκες, θα πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να ευθυγραμμίζουν την νομοθεσία τους. Αναφερθήκατε και στο πρόβλημα εφαρμογής. Ε, σαν να παλινοδεί δηλαδή η νομοθεσία μερικέ φορέ. Δεν θα το έλεγα αυτό. Απλώ είναι πιο, όλο και πιο δύσκολη η εφαρμογή τη ε, οδηγίας. Ωραία, καλά είναι τα, ε, τα θεωρητικά και οι νομοθετικές διατάξεις και καλή νομοθεσία. Αν δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στα θύματα, τότε προς τι η καλή νομοθεσία. Υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής και αναφέρθηκε και το θέμα του κόστους. Δεν γίνεται καμία επένδυση για να ε, καταρτιστούν οι δικηγόροι και οι δικαστές στις αρχές κατά των διακρίσεων και στην αντιμετώπιση των υποθέσεων διακρίσεων. Σε μερικές χώρες δεν αναφέρεται καν το θέμα ε, των διακρίσεων στο βιογραφικό ενός δικαστή ή ενός δικηγόρου. Πολλές φορές και οι δικαστές και οι δικηγόροι είναι άσχετοι με θέματα διακρίσεων. Οπότε θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις ε, και συνοδευτικά μέτρα. Γιατί η νομοθεσία δεν είναι το παν. Χρειαζόμαστε και συνοδευτικά μέτρα. Δεν μπορούμε να τα απειλήσουμε όλα νομοθετικέ διατάξει. Χρειαζόμαστε και μέτρα πολιτική και συνοδευτικά μέτρα για να ε, υλοποιήσουμε κάτι που προ στιγμή δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί από την νομοθεσία ή δεν καλύπτεται από την νομοθεσία. Σα ευχαριστώ. Περιμένουμε τώρα το σχόλιο και τον εμπειρογνωμόνων μα. Ο κύριο Δημητρακόπουλο πρώτα. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι δεν νομίζω ότι το επιχείρημα κόστος θα πρέπει να αναφέρεται σε μια συζήτηση για τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κάποιος πάντως το επικαλεστεί παρόλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχουν ήδη σαφή τεκμήρια και αποδείξεις από διάφορους τομείς. Γιατί στις δεκαετίες του 80 και του 90 έγιναν κάποιοι υπολογισμοί για την ε, θεσμοθέτηση, θεσμοποίηση όσων έχουν ε, νοητικές ε, καθυστερήσεις ή νοητικά προβλήματα είναι οι νοητικές αναπηρίες. Φάνηκε τότε ότι το κόστος ε, ε, μεγάλης εμβέλειας θεσμών ήταν πολύ σημαντικό. Υπάρχουν λοιπόν ε, ε στοιχεία ποσοτικά για το κόστος ε, διατάξεων ε, κατά των διακρίσεων. Επίσης υπάρχουν κάποια ευρύτερα θέματα που θίξατε και που δεν ε, συνοδεύονται ίσως από στοιχεία ή δεν τεκμηρώνονται με στοιχεία, αλλά συζητούνται σε μια πολιτική συζήτηση. Τι χάνουμε όταν ε, ε, υφίστανται άμεσες ή άμεσες διακρίσεις κάποιοι άνθρωποι που παρά τα προσόντα που έχουν δεν ε, μπορούν να βρουν τη θέση που τους αξίζει. Ένα Στίβεν Χόκινς με τα τεράστια προσόντα και τις δεξιότητες και την ε, ιδιοφία του, σκεφτείτε, παρά την, ε, και λόγω της αναπηρίας του, δεν είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει το δυναμικό. Τι θα έχανε η κοινωνία μας από αυτό. Ο κύριος Μάλινοφ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δημητρακόπουλο για ένα στοιχείο που μας έδωσε που μας ε, φέρνει και στο μεθοδολογικό ζήτημα. Είπατε ότι η πιο συνηθισμένη διάκριση είναι η διάκριση λόγω ηλικία. Το πιστεύω και εγώ. Αλλά μήπω είναι παραπλανητικό αυτό το στοιχείο. Γιατί όλοι γερνάμε αργά γρήγορα. Και ε, νομίζω ότι οι ηλικιωμένοι είναι όντως ε, θύματα διάκρισης. Αλλά νομίζω ότι στη δική μου πατρίδα η χειρότερη διάκριση δεν είναι, είναι λόγω ηλικίας. Αν κάνει κανένα δημοσκοπήσεις, ίσως ε, τα στοιχεία δείξουν ε, ότι ε, η πιο σοβαρή διάκριση είναι λόγω ηλικία, αλλά είναι επειδή υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που το επικαλούνται. Νομίζω είναι παραπλανητικό όμως να το αναφέρουμε ως πρωτοχικό στόχο διάκρισης. Έχετε εσείς κάποια στοιχεία ε, γιατί διάφορα είδη διακρίσεων, γιατί άλλες διακρίσεις είναι πιο έντονες στις ε, πρώην ανατολικές χώρες και άλλες στις ε, δυτικές χώρες. Γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν μακροχρόνια παράδοση με τέτοιου είδους ομοθετικές διατάξεις και άλλες που είναι πολύ πιο νέες σε κάτι τέτοιο. Μερικές χώρες θα χρειαστεί να μειώσουν τις προδιαγραφές τους λόγω της ε, πιθανής έγκριση αυτής της οδηγίας, γιατί αν ε, χρειαστεί κάτι τέτοιο, τότε λογικά είναι να είναι μερικές χώρες κατά. Ερωτώ, ποιες κρατικές νομοθεσίες είναι πολύ πιο φιλόδοξες ε, και προβλέπουν πολύ καλύτερες συνθήκες από ότι η ενδεχόμενη οδηγία αυτή αν εγκριθεί. Άλλα σχόλια παρακαλώ από τους εμπειρογνώμονες για τα σχόλια του κ. Μαλινόφ. Όχι, καμία χώρα δεν θα αναγκαστεί να μειώσει το επίπεδο προστασίας. Αναφέρθηκε και το θέμα το φιλετικών διακρίσεων. Χώρες ε, που έχουν ανώτερο επίπεδο προστασίας, όπως συνέβη και με, τη με την οδηγία κατά το φιλετικών διακρίσεων, μπορεί να το κρατήσουν. Δεν είναι επιχείρημα αυτό να πούν χώρε ότι εμεί έχουμε πολύ καλύτερο επίπεδο προστασία. Αν ε, εγκρίνουμε την οδηγία, θα πρέπει να το υποβαθμίσουμε. Δεν ευσταθεί αυτό το επιχείρημα, γιατί καμία χώρα δεν πρόκειται να ε, υποχρεωθεί να, υποτιμήσει, να υποβαθμίσει το επίπεδο προστασίας της. Άλλα σχόλια δεν βλέπω. Οπότε περνάμε στο τρίτο πάνελ. Α, α, ρώτησα αν ήθελε κανείς να κάνει σχόλιο. Έχετε το λόγο κύριε Δημητρακόπουλε. Να απαντήσω στα σχόλια που ακούστηκαν. Το θέμα της ηλικία. Όταν μιλάμε για ηλικία, δεν μιλάμε μόνο για ηλικιωμένους, μιλάμε και για τα παιδιά και για τους νέους. Δεύτερον, η ηλικία επηρεάζει και τις ερωτικές μειονότητες όπου οι, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά αυτών, κάποιων εθνικοτήτων μπορεί να υποφέρουν περισσότερο. Υπάρχει ε, διάφοροι τρόποι μέτρησης. Το Ευρωβαρόμετρο ρωτά τα, τους πολίτες ε, πόσο σημαντική είναι η διάκριση στον α τομέα. Ένα άλλο έρευνα, αυτό που κάνουμε εμεί, είναι ότι ερωτάμε ομάδε συγκεκριμένε σχετικά με την εμπειρία του πάνω στα θέματα διακρίσεων. Όταν αναβαίνουμε στο Ευρωβαρόμετρο, πρόκειται για την αντίληψη τη κοινή γνώμη για το ποιο ε, επηρεάζεται περισσότερο. Όταν κάνουμε εμείς ε, τις έρευνές μας ε, βλέπουμε ότι η ηλικία είναι σημαντικός παράγων που διατρέχει και όλες τις ηλικίε ε, και όλα τα φύλλα. Ωραία. <clears throat> Είμαστε έτοιμοι τώρα να περάσουμε στο τρίτο πάνελ. τρίτο τμήμα λοιπόν της ε, σημερινής μας συνεδρίασης ε, σχετικά με την αντιμετώπιση των ε, εμποδίων για την, σε θέματα ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δράσεις που θα πρέπει να αναλυφθούν να, για να απεμπλακεί η οδηγία την οποία εξετάσαμε τώρα. Και τώρα λοιπόν εξετάζουμε τα εμπόδια περιλαμβανομένου και του κόστου της δαπάνης. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε να έρθουν εδώ στο Προεδρείο ο κύριο Τομπίας Μπιούλινγκ Μαϊζίβεν ε, πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριε Τομπίας Μιούλεν Σίφεν διευθυντής ε, για την ισότητα τον κύριο Ζιώργιο Φιντεβίτε πρόεδρο της Equinot, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τους Φορείς Ισότητας και κάποιους εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων για θέματα διακρίσεων. Age, Platform Europe, την κυρία Αν Σοφή Παρό, παρακαλώ, προσέλθετε. Disability, EDF, κυρία Καρλότα Μπεζότσι σεξουαλικός προσανατολισμός ILGI, κύριο Γκρέγ Καρνέσκι και Religion and Belief, ENAR, κύριο Μάικλ Μικαέλα, θέλετε, Πρίβοτ. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από προσκεκλημένους οι οποίοι θα μας μιλήσουν για τα θέματα και για τις οργανώσεις που εκπροσωπούν. Θα έχουμε και στο τέλος 30 λεπτά στη διάθεσή μας. Για ερωταποκρίσεις, το λόγο έχει ο κύριος Τομπίας Μιουλεσίφεν για 10 λεπτά κύριε Τομπίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε εκ νέου να μιλήσουμε. Ακούσαμε σήμερα την παρουσίαση από τον Διευθυντή μου για ένα θέμα πιο πολιτικής φύσης και αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω αυτό το δεκάλεπτο που έχω διευθύνει μου είναι να αναφερθώ ποια είναι τα επίμεχα σημεία τα οποία συζητώνται στην ομάδα του Συμβουλίου Ακούσαμε φωνές υπέρ της διαφάνειας και θα σας μιλήσουμε για το τι συζητήσαμε τα τελευταία 3,5 χρόνια στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και να σας πω που έγκυται τα πρώτα θα σας μιλήσω για πολιτικά θέματα αλλά για τεχνικής φύσης ζητήματα τα οποία αποτελούν τμήμα των εργασιών. Σίγουρα θα γνωρίζετε την βασική δομή της πρότασης. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα. Ε, η θρησκεία, η του Ανατολισμό, η ηλικία και οι πεπιθήσεις, ε, αυτά είναι θέματα τα οποία δεν έχουν ακόμα αμφισβητηθεί στην ομάδα εργασία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να δουλεύουμε μια πρόταση που καλύπτει αυτά τα τέσσερα πεδία προστασίας και το ε, περιεχόμενο υπάρχουν δύο τμήματα το κομμάτι που αφορά τη μη διακρίσεις που είναι παρόμοια με την οδηγία περί ρατσισμού και, αφορά, και το δεύτερο κομμάτι αφορά τα θέματα των ατόμων με αναπηρία, δηλαδή την πρόσβαση και την ε, προσαρμογή. Θα θίξω τα διάφορα ζητήματα τα οποία μας απασχολήσει μέχρι τώρα. Ένα τα πιο σημαντικά είναι το πεδίο της οδηγίας διότι όπως γνωρίζετε καλύπτει τρεις τομείς, την πρόσβαση σε υπηρεσίες ε, και αγαθά, κάτι που αγοράζεται καθημερινά, αλλά συμπεριλαμβάνει και το θέμα της στέγασης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ε, δεύτερο είναι η κοινωνική προστασία που αφορά και την ε, περίθαλψη και το τρίτο είναι η εκπαίδευση, η παιδεία. Και εδώ έχουμε το ζήτημα ότι κάποια κρατημέλη ότι θεωρούν πως υπάρχει αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα για θέματα προστασίας. Ε, αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να αποκλειστούν από την και που θα αφορούν ε, την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε. Ε, έχουν γίνει διάφορε προτάσει, ειδικά για να διευκρινιστεί ότι η οργάνωση και η χρηματοδότηση τη κοινωνική προστασία και τη εκπαίδευση αφορά, είναι αποκλειστική αρμοδία των κρατών μελών. Όταν μιλάμε για πρόσβαση στα ωφέλη στι συγκεκριμένε ε, υπηρεσίε, τότε αυτά θα πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία. Πάντα φυσικά σε θέματα που αφορούν ε, στην προστασία. Ε, τώρα κάτι άλλο είναι ότι θα πρέπει να ε, δούμε σε ποιους υπηρεσίες και αγαθά εφαρμόζεται. Θα πρέπει να αφορά στα άτομα όταν ασκούν την οικονομική και εμπορική δραστηριότητα. Αυτό δεν είναι ένα ουσιαστικό κριτήριο και πιο σημαντικό κριτήριο είναι να μην υπάρχει ανάμειξη στην προσωπική και οικογενειακή ζωή. Δύο περιπτώσει που δεν θα εφαρμόζει η οδηγία είναι πρώτον αν τα αγαθά και υπηρεσίε δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό, δηλαδή εάν αγοράτε το, πουλάτε μάλλον το αυτοκίνητό σα σε κάποιον φίλον, αυτή η, συναλλαγή δεν θα, σε αυτή δεν θα εφαρμόζεται η οδηγία, αλλά εάν το αναφέρετε αυτό το θέμα στο διαδίκτυο, τότε θα καλύπτεται. Και επίση δεν θα καλύπτεται εάν οι συναλλαγέ γίνονται στο πλαίσιο τη οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, εάν νοικιάζετε ένα δωμάτιο στο διαμέρισμά σα ή αν έχετε κάποιον ε, φοιτητή ο οποίο μένει κατοικεί στο σπίτι σα ε, για λόγους γλωσσικούς ε, δεν θα καλύπτεται. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί είναι το θέμα της ηλικία. Υπάρχουν ποικίλα όρια ηλικία. Όταν μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση, για εκπαίδευση, παιδεία, υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες που αφορούν στην ηλικία. Έχετε κάποια ε, ωφέλη αν έχετε κάποια ηλικία, αν ξεπεράσετε δεν τα έχετε πλέον η Τούμπαλιν. Εάν ε, λάβετε υπόψη την ε, οδηγία περί εργασίας, βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχουν παιδεία για ε, εφαρμογή για ε, ε, διακρίσεων λόγω ηλικία. Θα χρησιμοποιήσω τώρα νομική ορολογία, η διαφορετική μεταχείριση για λόγους ηλικίας μπορεί να δικαιολογηθεί εάν ο στόχο ο οποίο πρέπει να επιτευχθεί είναι σύμφωνο με την αναλογικότητα. Υπάρχει ένα θέμα αναλογικότητα. Πρέπει να υπάρχει κάποιο, μπορεί να υπάρχει κάποιο όριο ηλικία και διάκριση, αλλά πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα. Υπάρχει λοιπόν μια ζήτηση στο Συμβούλιο σχετικά με το πώς ε, θα πρέπει να προληφθούν ε, σοβαρά προβλήματα. Μια επιλογή θα ήταν το, ε, τεκμήριο της ηλικία ε, το οποίο μπορεί να είναι δικαιολογημένο και ένα δεύτερο τρόπο θα ήταν ο αποκλεισμό ε, κάποιες ε, ηλικία από κάποιες περιπτώσεις όπως κοινωνική προστασία κλπ. Αυτά είναι θέματα που εξετάζουν Ένα τρίτο ζήτημα οικονομικές υπηρεσίε και ειδικά το ζήτημα της ασφάλειας το οποίο έχει γίνει καθημερινή συζήτηση, γίνει καθημερινή συζήτηση μετά από την απόφαση για την υπόθεση τεστ ΑΣΑ. Και έχουμε μια εξαίρεση στο κείμενο που αναφέρει ότι η διαφορετική ε, αντιμετώπιση με βάση την ηλικία μπορεί να δικαιολογηθεί εάν ε, συνυπολογιστεί και ο κίνδυνος ε, που συνδέεται με την ηλικία. Αλλά θεωρείτε ότι αυτή η εξαίρεση μπορεί να ε, προσβληθεί σύμφωνα με την απόφαση την υπόθεση τεστ ΑΣΑ. η ασφάλεια ζωής ε, μπορεί να μην ισχύσει αν, ε, αν υπόψη την ηλικία. Όλοι μπορούν να το κατανοήσουν αυτό. Ε, το θέμα συζητείται πως ε, μπορεί να γίνει κάποια κράτη-μέλη είναι υπέρ της ε, εξαίρεσης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών άλλα κράτη είναι κατά αλλά η εργασία μέχρι τώρα εστιάζεται στο να ενδυναμωθεί το κείμενο και να περιορίσουν τον κίνδυνο νομικής προσβολής της εξαίρεσης. Το τέταρτο ζήτημα είναι η έννοια της διάκρισης. Τι σημαίνει διάκριση, τι εννοούμε. Αυτό που δεν είναι προβληματικό και δεν το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα είναι ο ορισμός της άμεσης έμεσης διάκρισης. κάποια κράτη έχουν αποκτήσει εμπειρία με βάση τις προηγούμενες οδηγίες. Αυτό το οποίο όμως είναι αντιφατικό είναι ο ο ορισμός της παρενόχλησης και διεξάγεται συζήτηση και με το πόσο είναι ιδιαίτερα ευρύς παρενόχληση μπορεί να έχουμε μόνο όταν είναι επαναλαμβανόμενη. Δεν μπορεί να είναι μία, μία και έξω. Πρέπει να υπάρχει επανάληψη και να είναι αρκετά, αλλά φυσικά μόνο αν είναι αρκετά σοβαρή η παρενόχληση που διεξάγεται άπαξ, μόνο τότε μπορεί να θεωρηθεί πραγματική παρενόχληση. Διαφορετικά θα πρέπει να είναι μια παρενόχληση η οποία να επαναλαμβάνεται. Ένα άλλο ζήτημα είναι ε, στις ε, ε, διάκρισεις με η διάκριση by association. Αλλά τότε με την έκθεση Buitenweg είχε υπολυθεί μια τροπολογία η οποία έγινε δεκτή, αλλά το ζήτημα είναι πώς θα πρέπει να οριστεί, διότι μπορεί να ε, πέσουμε σε ένα πολύ ευρύ ορισμό. Και τέλος, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, το οποίο μας απασχολεί στο Συμβούλιο, είναι το δεύτερο τμήμα της ε, πρότασης, ε, τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία το ζήτημα της προσαρμογής, της προσβασιμότητας. Η προσβασιμότητα ξέρετε ότι είναι γενικά προληπτικά μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να βρείτε τα εμπόδια και να τα αφαιρέσετε, να τα εξελίψετε, ενώ η προσαρμογή είναι μέτρα ad hoc, κατά περίσταση. Οπότε πώς μπορείτε να κάνετε κάποιες διευθετήσεις προκειμένου ο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση όλα αυτά θεωρούνται ότι δεν έχουν ε, οριστεί με τρόπο απτό και συγκεκριμένο. Γιατί είδου ε, αναπηρία καλύπτουμε, δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειε στο κείμενο γιατί κάνουμε το τι θα πρέπει να κάνετε για άτομα που είναι σε αμαξίδιο, για άτομα ε, του τυφλού κλπ. Υπάρχει και το θέμα της σύμβασης του ΟΗΕ, διότι θα, υπήρχε, θα ήταν καλό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει μια παρόμοια προσέγγιση με αυτήν όλα τα κρατημέλη. Θα πρέπει να την ε, εφαρμόσουν να είναι λοιπόν κάποιες προτάσεις, κάποιες συστάσεις επί του κειμένου. Προτείναμε λοιπόν ένα μεγαλύτερο χρονικό όριο για να λάβουμε υπόψη και τον κύκλο ζωής των κτηρίων. Δεν θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά μέσα σε δύο-τρία έτη που είναι συνήθις χρόνο για την υλοποίηση εφαρμογή της οδηγίας. Υπάρχουν και συζητήσεις πολυτεχνικού χαρακτήρα σχετικά με τη στέγαση, πώς θα υπάρχει προσαρμογικότητα και ευλογή προσαρμογή σε ένα, για ένα διαμέρισμα προκειμένου αυτό να καταστεί προσβάσιμο. Συζητείται επίσης και το θέμα του της αναλογικότητας ε, του βάρους, του άχθους είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε και στο παρελθόν αλλά είναι μια αξιολόγηση κατά περίπτωση ε, διευκρινίσαμε ότι στη συζήτηση ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, είναι η αξιολόγηση αυτού του περαιτέρω βάρους, περαιτέρω φόρτου. Τώρα, ε, η ασφάλεια δικαίου είναι ένα γεγονός, αλλά ε, δεν μπορούμε να ε, διευθυντήσουμε όλα τα ζητήματα μέσα σε ένα νομοθέτημα. Υπάρχουν και ίσονο σημασία ε, ζητήματα. Υπάρχουν και κάποια άλλα όπως το ζήτημα του βάρους απόδειξης, θετική δράση, χρηματοποίηση και για τους φορείς ισότητας. Αυτά ήθελα να πω ως εισαγωγή για να γνωρίζετε τι συζητάμε στην ομάδα του Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε κύριε Μίλεν Ζήφεν. Περνάμε στο δεύτερο εμπειρογνώμονά μας, τον κύριο Γιώζεφ Ντεβίτε, τον πρόεδρο της ΕΚΟΙΝΕΤ, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων Ισότητας, για 10 λεπτά. Περιμένουμε την παρουσίασή σας κύριε Ντεβίτε. Έχω μια παρουσίαση με PowerPoint. Έχω, θα αρχίσω μια διαφάνεια, θα τελειώσω μια διαφάνεια και έχω μόνο έξι διαφάνειες συνολικά. Ελπίζω να λειτουργεί το μηχάνημα εδώ. Just a second. Let's see if it can be meant. Δεν ξέρω, τι διακρίσεις είναι αυτές. Λόγω ηλικίας μήπως ή λόγω φίλου. Όχι, όχι, δεν θα κάνω τις διακρίσεις εμείς. Καταρχήν η αποστολή της ΕΚΟΙΝΕΤ. ΕΚΟΙΝΕΤ είναι το δίκτυο φορέων ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να επιτρέψουμε στα, στους φορείς ισότητας να επιτύχουν και να ασκήσουν το πλήρες δυναμικό τους διατηρώντας και αναπτύσσοντας μια δικτύωση μεταξύ τους και μια πλατφόρμα φορέων ισότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η πολύ απλή αποστολή της Equinet, του Equinet μάλλον του δικτύου. Έχουμε φορείς ισότητας ε, γιατί και οι οδηγίες ε, ε, κατά των φυλετικών διακρίσεων και υπέρ τη ισότητα των φύλων προβλέπουν υποχρεωτικά σύσταση τέτοιων φορέων ισότητα ε, από τα κράτη-μέλη προκειμένου να παράσχουν αρρωγή στα θύματα της, ε, των διακρίσεων, να καταρτίζουν εκθέσει και μελέτε για θέματα διακρίσεων, να υποβάλουν συστάσεις για θέματα διακρίσεων και να ανταλλάσσουν πληροφορίε με ευρωπαϊκά όργανα. Ε, επίσης ε, να συμβάλλουν σε μια φύπνιση, στην καλών πρακτικών, είναι και αυτά αποστολές των φορέων ισότητα. Το δίκτυό μας, το Equinet, ε, ξεκίνησε το 2003. Οι πρώτε επαφέ ξεκίνησε το 2003, η επίσημη σύσταση το 2007. Έχουμε 27 φορεί ισότητα στις 27 χώρε μέλη. Και Φυσικά ασχολούμαστε με τις οδηγίες ε, κατά το φυλετικό διακρίσιο και υπέρ της ισότητας των φύλων. Βέβαια, ε, ασχολούμαστε και με την οδηγία ε, που αφορά διακρίσεις του, για τους τέσσερις λόγους που εξετάζουμε και σήμερα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των φορέων ισότητας στα κράτη-μέλη και το μέγεθός τους και η εντολή τους, οι λόγοι των διακρίσεων, η δομή και η εμπειρία τους είναι διαφορετικά. Αλλά αυτό είναι και το καλό με το δίκτυο. Ο πλούτο του δικτύου είναι ότι επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να αξιοποιήσουμε όλοι τις εμπειρίες και να υποφεληθούμε από τα καλά παραδείγματα. Έχουμε 34 μέλη είπαμε, στο δίκτυό μας, 27 είναι χώρες μέλη, 34 αφορούν ε, τις φιλετικές και θεωρητικές ακρίσεις, για 32 το φύλλο, 31 πίστη θρησκεία, 30 ηλικία, 30 ε, γενετήσιο προσανατολισμό και 29 ε, αναπηρία. Αυτή είναι η πρωταρχική λόγη διακρίσεων. Ποιες είναι, ποια είναι η προσθεθέμενη αξία των φορέων ισότητας σε αυτή τη συζήτηση για τη νέα οριζόντια οδηγία. Ε, ήδη το 2008 δημοσιεύσαμε μία γνωμοδότηση με τίτλο «Πέραν της αγοράς εργασίας». Όπως σας είπα, μας είπε και η κυρία Σοπέν ότι 20 κράτη-μέλη έχουν νομοθεσίες που ξεπερνούν ε, την, ε, το χώρο της απασχόλησης ε, για τους τέσσερις λόγους. Και ε, το Βέλγιο έχει ένα φορέα ε, ισότητας που αφορά τις, ε, τα αγαθά και τις υπηρεσίες για αυτούς τους τέσσερις λόγους. Ηλικία, ανα, αναπηρία, γενετήσιο προσανατολισμό και θρησκεία. Θα σας δώσω σε λίγο μερικά παραδείγματα για τους λόγους που καλύπτονται. Έχουμε περιπτώσεις διακρίσεων σε αγαθά και υπηρεσίες. Όπως είπα και προηγουμένως, στόχος του ΕΚΟΝΕΤ είναι να ενημερώνουμε και τους δικαστές για την ύπαρξη νομοθεσίας. Μερικές φορές βέβαια είναι επέσχυρο και τέτοιο, αλλά μας εντυπωσιάζει μερικές φορές η άγνοια των δικαστών. Βέβαια είναι σχετικά πρόσφατες αυτές οι νομοθετικές διατάξεις το Βέλγιο το 2003, αλλά πολλές φορές οι, δικαστές δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Όταν βλέπουμε από τη μια την απασχόληση και από την άλλη τα αγαθά και τις υπηρεσίες, διαπιστώνουμε το 2011 ε, στη, στη βελγική περίπτωση, είχα, στο βελγικό φορέα ισότητα, είχαμε περισσότερε περιπτώσει διακρίσεων στα αγαθά και τι υπηρεσίε από ό,τι στην απασχόληση. Επίση, ε, το δίκτυό μα ε, ασχολείται και με θέματα διακρίσεων λόγω ηλικία. Θα μα πει αργότερα τι γίνεται ο συνάδελφο με το έτσι. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Έτος για την ενεργό και διαπιστώνουμε ότι οι διακρίσεις λόγω ηλικία υπάρχουν όχι μόνο στην απασχόληση αλλά και στα αγαθά και τις υπηρεσίε. Από την εμπειρία μα από του φορεί ισότητα, ε, διαπιστώνουμε ότι όταν μιλούμε για απασχόληση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Ακούσαμε ένα παράδειγμα. Πώ μπορεί κανεί να ανεβεί σε ένα τρένο, να επιβεβαστεί σε ένα λεωφορείο, ακόμη και να πάρει ταξί. Είχαμε ένα ρεπορτάζ ενό βελγικού καναλιού ε, για το πώς μπορούν να, ε, να μπουν σε ταξί τυφλοί που χρειάζονται σκύλο συνοδό. Είχαν πρόβλημα ακόμη και να μπουν σε ταξί, στο Βέλγιο, κάτι που είναι απαράδεκτο. Αν κανείς θέλει να έχει απασχόληση και να κερδίζει ένα μισθό, θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε για να μπορεί να βρει μια δουλειά και να έχει και μισθό. Και μετά για να ξοδέψει το μισθό του πρέπει να έχει πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε. Γιατί αυτό είναι το περίεργο. Μερικέ φορέ κάποιο που έχει μισθό δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι εξαιτία των διακρίσεων ε, και των προβλημάτων στην πρόσβαση στο δανεισμό. Εσεί είστε τυχεροί, γιατί στι 12.30 στη διακοπή μπορείτε να πάτε και να γευματίσετε και δεν θα σα κλείσει κανεί την πόρτα στο εστιατόριο επειδή είστε ομοφυλόφιλο ή είστε επειδή πολύ νέο, πολύ γέρο ή επειδή είστε ανάπηρο. Με βάση τη βελική νομοθεσία, διακρίσει ε, απαγορεύονται όχι μόνο λόγω φίλου και φιλής, αλλά και λόγω αναπηρίας, γενετής προσανατολισμού, ηλικία, κάτι που δεν ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν υπάρχει αυτή η προστασία η διευρυμένη. Και είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές να εξηγήσουμε γιατί ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί μπορεί κανείς να, μη, να, να στερηθεί την είσοδο σε ένα εστιατόριο ή να, την είσοδο σε ένα ξενοδοχείο λόγω αναπηρία, της αναπηρίας του. Οι φορείς ισότητας, όπως ο Βελγικός για παράδειγμα, ε, χαίρεται που δεν υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις στο Βέλγιο τουλάχιστον ε, και για φιλετικούς λόγους ή για λόγους φίλου αλλά και για τους υπόλοιπους τέσσερις λόγους. Θα είναι πολύ δύσκολο όμως να εξηγήσει ένας φορέας ισότητας ότι δεν υπάρχει αυτή η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων σε ό,τι αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Ακούσαμε πολλές φορές την παράκληση. Εξηγήστε μας γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Ποια είναι η εξήγηση λοιπόν γιατί ορισμένες χώρες έχουν περισσότερη προστασία και άλλες όχι. Γιατί δεν υπάρχει μια κοινοτική οδηγία που να εξασφαλίζει αυτή την προστασία. Τώρα, υπέρβαση των εμποδίων. Εμείς παράσχουμε αρρωγή, παρέχουμε αρρωγή και στα θύματα. Και μάλιστα και για θέματα αγαθών και υπηρεσιών. Βρίσκουμε συγκεκριμένες λύσεις. Μερικές φορέ οι άνθρωποι είναι πανικόβλητοι και φοβισμένοι. Λέει τι θα γίνει με την οδηγία, θα καταιγιστούμε από παράπονα. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων των διακρίσεων είναι πολύ λογικοί άνθρωποι. Λύση απλώ θέλουν. Θέλουν απλώ να καταλάβουν το πρόβλημα, να διαπραγματευτούν και οι αντιδικίες είναι πολύ λίγες. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει αντιδικία, δεν θέλει διαμάχη στο δικαστήριο, λύση θέλει. Αλλά όταν ο νόμος δεν προβλέπει λύση, φυσικά θα προσφύγουν ε, και θα αντιδικήσουν. Αλλά γενικώ ο κόσμος είναι λογικός, είναι Αναφέρθηκε και ο λόγος ε, του CPRD, της Επιτροπής Προστασίας Δικαιωμάτων Αναπήρων, Πώς εξηγείται ότι υπάρχει συνθήκη του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων αναπήρων και δεν έχουμε μια τέτοια οδηγία που να ε, εφαρμόζει αυτή την προστασία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας εξηγήσουμε λοιπόν και συζητήσουμε στην Ευρώπη πώς θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συνθήκη, τη σύμβαση αυτή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αναπήρων. Τώρα, η ιεράρχηση των λόγων, αλλά και η ιεράρχηση της προστασίας. Υπάρχει μία ασυμβατότητα και εδώ και μία συνέπεια. Και αναφέρθηκε και η ελευθερία διακίνησης. Όταν κανείς πηγαίνει σε μια άλλη χώρα που πραγματικά δεν μπορεί να γευματίσει ένα εστιατόριο ενώ στο Βέλγιο μπορεί, πώς θα το εξηγήσουμε αυτό αν υφίσταται διακρίσεις λόγω ηλικίας, γενετήσεων ανατολισμό, αναπηρίας κτλ. Και τέλος μιλήσαμε για το κόστος. Το κόστος της οδηγίας ή το κόστος της διάκρισης. Πολλές μελέτες έγιναν και πολλές έρευνες που έδειξαν το κόστος της ε, διάκρισης. Υπάρχει κόστος και από την εφαρμογή των διακρίσεων. Για παράδειγμα, υπάρχει πρόβλημα στην πρόσβαση στην απασχόληση. Αν δεν έχει κανεί ε, δουλειά όμω, δεν θα έχει πρόσβαση και στα αγαθά και τις υπηρεσίες. Οπότε το κόστος της διάκρισης θα είναι τεράστιο και στο Βέλγιο είχαμε περιπτώσει ακριβώ επειδή κάποιο δεν μπόρεσε να βρει δουλειά, δεν μπόρεσε να αγοράσει ένα αξιοπρεπές σπίτι, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε. Αν σα ενδιαφέρει λοιπόν η απασχόληση, ε, υιοθετήστε και την οδηγία για τα αγαθά και τι υπηρεσίε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεβίτε. Α ακούσουμε τώρα του εκπροσώπου ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων όπω ανακοινώθηκαν. Ξεκινάμε ε, από την ε, πλατφόρμα της Ευρώπης για την ηλικία. Η κυρία Άνσοφη Πάουντ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ε, μην θεωρήσετε ότι οι διακρίσεις λόγω ηλικία είναι ε, σημαντικότερες από ε, διακρίσεις για άλλους λόγους. Ε, Ακούσαμε διάφορα πράγματα. Έχουν ξεκινήσει κάποιες ε, προσπάθειες ε, επί Πολωνικής Προεδρίας ε, και τώρα δίδεται συνέχεια από τη Δανέζικη Προεδρία. Νομίζω ότι ο λόγος που αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στι διακρίσει λογοηλικίας δεν είναι ότι είναι πιο σημαντικές διακρίσει αυτές, αλλά είναι νέα έννοια για πολλά κράτη-μέλη. Είναι κάτι το οποίο πριν δεν το αναφέραμε καν. Και όλα ξεκίνησαν με την ε, οδηγία περί απασχόλησης ε, που ε, ξεκίνησε με την έννοια της, των διακρίσεων λόγω ηλικίας στην απασχόληση. Είναι πάντως ένα φαινόμενο που υπάρχει. Σχεδόν παντού υπάρχουν, γίνονται αναφορές σε, στην ηλικία στις ε, κοινωνικές υπηρεσίες, ε, στην εκπαίδευση. Ε, δεν λέμε ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα όρια ηλικίας. Αναγνωριζόμαστε ότι η κοινωνία μας είναι οργανωμένη γύρω από τον κύκλο ζωής. Αυτό το αναγνωρίζουμε, ούτε λέμε ότι είναι λάθος. Ξέρουμε όμως από τις εμπειρίες που έχουμε από τα μέλη μας και από τη δουλειά που έχει γίνει όχι μόνο από μας αλλά και από άλλους εμπειρογνώμονες ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου η ηλικία χρησιμοποιείται με καταχρηστικό τρόπο. Να σας εξηγήσω γιατί πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη αυτή η οδηγία. Ε, ζούμε σε ένα πλαίσιο ε, γύρανσης του πληθυσμού ε, Έχουμε όμως και την εντύπωση ότι όσο πιο γρήγορα γερνάμε, τόσο λιγότερο προσαρμοσμένη είναι η κοινωνία μας ε, στη γύρανση και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Έχουμε όρια ηλικίας ε, τα οποία δεν, μπορεί, ε, δεν έχουν πια νόημα. Μπορεί να είχαν νόημα πριν λίγο καιρό, αλλά όχι πια. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η νομοθεσία, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα κάποιων κρατών μελών, που προχώρησαν ε, πέρα από τα όσα απαιτούνται από την απλή ε, μεταφορά τι οδηγίε για την απασχόληση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με διαφορετικό τρόπο την ηλικία από ό,τι ε, ε την βλέπαμε στο παρελθόν. Και γι' αυτό ε, οι ανταποκρίσει στο ευρωβαρόμετρο όταν τους ρωτούν στο Ευρωβαρόμετρο ε, ποιος είναι ο πιο σοβαρός τρόπος ε, διακρίσεων που γίνεται, ε, η ηλικία βρίσκεται σε αρκετά υψηλή θέση. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Στην απασχόληση, οι διακρίσεις λόγω ηλικίας είναι πρόβλημα και για τους πολυνέους και για τους πολυμεγάλους. Αν δείτε τα ποσοστά απασχόλησης στις δύο αυτές ομάδες θα το διαπιστώσετε το ίδιο ή σε κάποιους τομείς της ζωής μας έξω από την απασχόληση. Πιο προβληματικό ε, είναι η πρόσβαση σε ε, χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπάρχει ειδικό άρθρο στην ε, οδηγία για τις διακρίσεις. Χρειαζόμαστε πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λόγω τρόπου που λειτουργεί η κοινωνία. Χρειαζόμαστε πρόσβαση στις, ασφάλεις, στις ασφαλίσεις, για παράδειγμα. Και Έχουμε βρει δύο διαφορετικές κατηγορίες χρηματοπιστωτικών ε, προϊόντων που παρουσιάζουν διαφορετικά προβλήματα. Κάποια ε, προϊόντα, για παράδειγμα ε, η ασφάλιση ταξιδίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπάρχει όριο ηλικίας. Ε, η δικαιολογία των ασφαλιστικών ε, επιχειρήσεων ε, είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος οι ηλικιωμένοι να χρειαστούν έκτακτη βοήθεια όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα από τη δική τους. Αυτό όμως δεν ισχύει εντός Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει συντονισμός των κοινωνικών υπηρεσιών, το οποίο σημαίνει ότι αν καλύπτεται κανείς στην πατρίδα του, καλύπτεται και στο εξωτερικό και αυτό καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση ε, στο, στην πατρίδα σας. Ε, αυτή λοιπόν είναι καταχρηστική χρήση ορίων ηλικίας και θα πρέπει να απαγορευτεί για να προωθηθεί και να διασφαλιστεί ε, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα ελεύθερη κινητικότητα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ισχύει λοιπόν αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολύ σαφή παραδείγματα. Μερικοί από εσά μπορεί να αμφισβητείτε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά είχαμε μια ασφαλιστική ε, ε, στην Ισπανία. Δεν μπορεί να αγοράσει κανεί ταξιδιωτική ασφάλιση αν είναι άνω των 65 ετών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το όριο είναι 70. Ε, μερικές φορές ε, είναι πολύ ψηλά τα τέλη για αυτούς άνω των 65 ε, ή σε μερικές περιπτώσεις δεν παρέχεται η ασφάλιση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν παρέχεται ασφαλιστική, ταξιδιωτική ασφάλιση άνω των 60. Μπορεί εσείς ως ευρωβουλευτές να έχετε ιδιαίτερες διατάξεις όταν ταξιδεύετε στις Βρυξέλλες αλλά τα δύο τρίτα των μελών μας ε, που ε, εκπροσωπούν ε, ενώσεις ηλικιωμένων σε όλη την Ευρώπη δεν μπορούν να έχουν ασφάλιση όταν ταξιδεύουν στις συναντήσεις μας. Υπάρχουν και τραπεζικά προϊόντα με όρια ηλικίας τα οποία μπορεί να φαίνονται πολύ λογικά από κάποια ε, άποψη. Για παράδειγμα, αν θέλει κανείς ασφάλεια ζωής όταν ε, είναι 98 ετών, ε, φυσικά ο κίνδυνο είναι τελείω διαφορετικό από ότι όταν είναι 25. Αλλά όταν θέλει να αγοράσει κανείς συμπληρωματική ασφάλιση υπάρχουν διακρίσεις. Ε, φυσικά οι πιο ηλικιωμένοι χρειάζονται περισσότερη περίθαλψη από ότι οι νεότεροι, αλλά το πρόβλημα αυτό δεν είναι πρόβλημα για ε, τις ασφαλιστικές εταιρείες, ε, διότι υπάρχει μια τάση σε όλη την Ευρώπη να βασιζόμαστε περισσότερο σε συμπληρωματική ασφάλιση για να διασφαλιστεί η επαρκής πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Αυτό σημαίνει ότι, όπως στη Γαλλία, οι ηλικιωμένοι πρέπει να πληρώσουν τεράστια ποσά για να έχουν συμπληρωματική ασφάλιση, ώστε ε, να μην ε, μπορούν να την πληρώσουν ε, στη στιγμή τη ζωή τους που τη χρειάζονται. Τέτοια κοινωνία θέλουμε. Αυτό είναι ερώτημα όχι για τους ασφαλιστές, είναι για αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική. Η στους ασφαλιστές δεν αρέσει ο κίνδυνος και δεν θέλουν ε, να καλύπτουν κινδύνους ε, που θα, ε, που θα εμφανιστούν κατά 100%. Και τέλος έχουμε το θέμα του κόστους, το οποίο συνδέεται με τις εύλογες προσαρμογές και την ανάγκη να οργανώσουμε την κοινωνία μας, ώστε να διασφαλίσουμε την ενεργογύρανση. Και από τη στιγμή που ε, δημιουργούμε ε, εμπόδια, εμποδίζουμε τον κόσμο να ε, εργαστεί και τους εμποδίζουμε να συμμετέχουν στην κοινωνία. Να σας δώσω το παράδειγμα κάποιων χωρών που έχουν επενδύσει σε ε, ε, περιβάλλοντα υποστήριξη. Στη Σουηδία και στη Δανία έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ε, απασχόλησης στους ηλικιωμένους. Έχουμε μεγαλύτερο ε, ποσοστό αποσχόληση γυναικών, διότι δεν χρειάζεται να φύγουν από την αγορά εργασία ε, για να φροντίσουν τα μέλη της οικογένειας. Ε, σίγουρα τα περιβάλλοντα υποστήριξης αποτελούν πολύ καλή επένδυση. Ελπίζουμε ότι η τεχνική πτυχή των εύλογων προσαρμογών και το πώς μπορεί να γίνει ε, πιο ε, ε, υποστηρικτικό το περιβάλλον για όλους μας, είτε είναι, έχει κανείς κάποια αναπηρία, είτε απλά γεννάει και χρειάζεται ένα πιο προστατευτικό περιβάλλον. Ελπίζουμε ότι θα λυθεί το θέμα αυτό, ώστε να στηρίξουν όλα τα κράτη-μέλη την οδηγία αυτή, την οποία χρειαζόμαστε πάρα πολύ. αλλά αξίζει τον κόπο να δούμε από επιχειρηματικής πλευράς ε, τις επενδύσεις σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, διότι τα κράτη-μέλη ε, πρέπει να θέσουν προτεραιότητες. Αλλά πιστέψτε με, τα κράτη-μέλη που έκαναν τέτοιες επενδύσεις, όπως για παράδειγμα η Σουηδία, είδαν ε, απότομη πτώση ε, στην ε, ε, ε, ε, στην απασχόληση των ηλικιωμένων κτλ. Όχι επειδή έχει βελτιωθεί η υγεία τους, αλλά επειδή το περιβάλλον του υποστηρίζει περισσότερο, οπότε οι, οι ηλικιωμένοι να μπορούν να είναι πιο ανεξάρτητοι και να μην επιβαρύνουν την κοινωνία. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα την κυρία Καρλώτα Πεζότσι που θα μας μιλήσει για τις αναπηρίες. Ευχαριστώ. Είμαι από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίες. Είναι μια οργάνωση που συνεργάζεται με εθνικές και ευρωπαϊκές οργανώσεις και που περιλαμβάνει τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Ιδρυθήκαμε το 1976 Ε, κατά πολέμη των διακρίσεων θέματα αναπηρίας ήταν ε, και συνεχίζει να είναι ο ουσιαστικός αγώνας μας. Το άρθρο 5 της συνθήκης ε, του Άμστερνταμ ήταν κάτι που μας απασχόλησε διότι την εποχή εκείνη. Θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε το ζήτημα των διακρίσεων και της αναπηρίας να θεωρείται ε, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας. Και ακούσαμε κάποια παραδείγματα προηγούμενα αναφορικά με τα θέμα της υλοποίησης της ε, νομοθεσίας ε, περί αποφυγής διακρίσεων Όπως και όλες οι μη κυβερνικές οργανώσεις που παρίστανται εδώ, εκφράσαμε την ικανοποίησή μας ότι υπήρξε μια νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, αλλά και την ε, θέμα της ε, αναπηρίας ε, είχαμε ξεκινήσει έναν αγώνα για να λάβουμε ένα εκατομμύριο υπογραφές το λεγόμενο One Million Disability Campaign. Τελικά ε, ικανοποιηθήκαμε από το γεγονός ότι η προσπάθειά μας ε, ευωδόθηκε, μπορέσαμε λοιπόν να προχωρήσουμε παρακάτω. Αλλά και κάποια από τα ζητήματα δεν μας ε, τα οποία αναφέρθηκαν και εδώ σε προηγούμενη, στην προηγούμενη συζήτηση, π.χ. ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα αναφορικά με τις υπηρεσίες ασφάλισης. Έχουμε κάτι πολύ πιο αδύναμο από το το οποίο θέλαμε ε, και θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης προσώπων με αναπηρία. Υπάρχει κάποια σύγχυση ανάμεσα στην πρόσβαση στην ε, παιδεία και την ειδική εκπαίδευση που δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται σε μια παρόμοια οδηγία, αλλά υπάρχουν και κάποια ζητήματα γύρω από το θέμα της πρόσβασης και μια σύγχυση που υπάρχει με την εύλογη προσαρμογή. Τώρα βρίσκω ότι έχουμε βαλτώσει σε επίπεδο Συμβουλίου και για μας αποτελεί ένα όνειρο αλλά και μια πραγματικότητα, μια ανάγκη συγγνώμη, να εφαρμοστεί οδηγία για άτομα με αναπηρία Τα άτομα με αναπηρία συχνά ε, είναι αόρατα στην κοινωνία μας. Ε, εντάξει, υπάρχει η σύμβαση, σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία. Πραγματικά αποτελεί έναν οδηγό, διότι υπάρχει υποχρέωση προς τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μια σειρά διατάξεων και ειδικά ε, μη διακρίσεις και την προσβασιμότητα που βρίσκονται στον πυρήνα της ε, σύμβαση. Υπάρχει και ένα άρθρο το οποίο είναι αρκετά ισχυρό και που συνδέει την προσβασιμότητα με την εύλογη προσαρμογή η οποία πάει πέρα από το όσο περιέχει η οδηγία και θα είχε νόημα να έχουμε μια οδηγία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι υπάρχουν κράτη που εφαρμόζουν ήδη σχετική νομοθεσία, αλλά υπάρχουν και άλλα κράτη τα οποία η νομοθεσία καλύπτει κάποιες μόνο πτυχές, δεν είναι συνεκτική η νομοθεσία τους και η δυσκολίες ε, συνεχίζουν να εφίστανται από τη στιγμή που δεν υπάρχει ε, μια κοινή οδηγία, μια κοινή νομοθεσία για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν των πολιτικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση διότι έχει προσυπογράψει τη σύμβαση, διότι ε, μην ξεχνάμε ότι 27-27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυρώσει την συμφωνία διεξάγεται μια συζήτηση αυτή την εποχή γύρω από το κόστος, από τις δαπάνες που θα προκύψουν. Επίσης ακούστηκε σήμερα ότι υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία που δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα ιδιαίτερο με το κόστος αλλά το ζήτημα της απασχολεί. Ακούστηκε ότι υπάρχει και το κόστος από τη μη εφαρμογή της ε, νομοθεσίας ε, π.χ. Ε, χωριστά συστήματα τα οποία ισχύουν. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα ειδικά σχολεία, για άτομα τα οποία δεν μπορούν να εργαστούν. Όλο αυτό φυσικά δημιουργεί περαιτέρω κόστος και θα θέλω να επανέλθω τώρα στο παράδειγμα που έδωσε ο κύριος Ντεουίτ σχετικά με την ε, βελγική νομοθεσία που καλύπτει ε, διακρίσεις σε αφορά την πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Αυτό ισχύει και στο ο Βασίλειο αλλά και στην νομοθεσία για την απασχόληση και δεν είδαμε ποτέ να χρεοκοπεί καμία επιχείρηση διότι πρόβλεψε να προσαρμόσει κατάλληλα τις εγκαταστάσεις της. Αυτές οι επιχειρήσεις ε, συνεχίζουν να λειτουργούν και αν ε, έπαψαν να δραστηριοποιούνται δεν οφείλεται σε μια δικαστική απόφαση επειδή δεν ε, φρόντισαν να παρέχουν εύλογες προσαρμογές. Ένα άλλο θέμα κλειδί το οποίο συζητείται στο Συμβούλιο και που χρειάζεται να διευκρινιστεί περαιτέρω αφορά την σύγχυση σε ε, θέματα προσβασιμότητας με την ευλογή προσαρμογή. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι χρήσιμη, κάποιες αλλαγές ε, έχουν γίνει και στο Συμβούλιο που βοήθησαν να διευκρινιστεί η ανάγκη ανταπόκριση σε ατομικές ε, προσωπικές ανάγκες αλλά και το δυσανάλογο άχθος που συνδέεται και που διαχωρίζει το ζήτημα της προδασιμότητας εκ των προτέρων ε, μέσω της κατάλληλης πρόβλεψης. Και εδώ πιστεύω ότι είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης ε, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και τώρα επανέρχομαι σε ένα σχόλιο που έγινε από την κοινωνική πλατφόρμα προηγούμενα να συνεχιστούν συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και να ακούσουμε εμπειρογνώμονες, ε, πως επίσης στην εμπειρία των μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων, να ανοιχθεί συζητήσεις ε, με κάποια, κάποιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, για θέματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ασφάλισης, που καλύπτουν και θέματα εκπαίδευσης, παιδείας, προσβασιμότητας και να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια δήματα που συζητούνται στο Συμβούλιο. Αυτές είναι κάποιες από τις πρακτικές λύσεις συναντήσεις σαν τη σημερινή που μπορεί να οργανώσει το Κοινοβούλιο και στο μέλλον είναι απόλυτα χρήσιμες για την επεμπλοκή της οδηγίας και για περαιτέρω συζητήσεις. Τέλος, να κάνω ένα σχόλιο για το θέμα της πολιτικής βούλησης. Εάν δούμε τις προσπάθειες που κάποιες <clears throat> αναπτυσσόμενες χώρες κάνουν προκειμένου να εφαρμόσουν την ε, σύμβαση του ΟΗΕ και την έλλειψη βούλησης ε, που παρατηρούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρώ ότι αυτό αποτελεί εδώ Η Ευρώπη λοιπόν δεν μπορεί να επικρίνει άλλα κράτη σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, τη στιγμή που δεν αναλαμβάνει τις, δικέ τις δικές της ευθύνες για θέματα καταπόλυψης διακρίσεων κλπ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα σε άλλη μια κυβερνητική οργάνωση, την ε, ILGA Europe, ε, διακρίσεις λόγω γενετήσου προσανατολισμού. Το λόγο κύριος Γκρέγκ Τσαρνέτσκι, ονομάζομαι Γκρέγκ Τσαρνέτσκι από την ILGA Europe τη διεθνή οργάνωση ε, LGBT, λεσβιών, ομοφιλοφίλων, αφιφιλοφίλων, ε, διαφιλικών, φιλομεταβατικών. Αν συγκρατήσετε τι σημαίνουν τα αρχικά μέχρι το τέλος της ακρόασης, ε, θα είμαι πολύ ε, ικανοποιημένος. Ανήκω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Elga Europe, θα ε, υιοθετήσω ένα διαφορετικό πρίσμα από αυτό των προλελισάντων των άλλων κυβερνητικών οργανώσεων ε, υπάρχει μεγάλη αντίσταση στην οδηγία αυτή και είναι διαφορετική η αντίσταση όταν μιλούμε για το γενετήσιο προσανατολισμό. Και το ανέκδοτο που μας ανέφερε ε, η κυρία Λούνατσεκ από τα Eurogames των ομοφιλοφίλων ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί η Γερμανία όντως είναι μία από τις χώρες που δεν είναι στο πλευρό μας γιατί αντιμάχονται ε, είναι μια από τις χώρες που αντιμάχεται τις οδηγίες. Βέβαια, για λόγους ε, αναπηρίας και όχι για λόγους γενετήσεων προσανατολισμού. Όντως, ε, δεδομένη της γενετήσεις ταυτότητας του κ. Βεστερβέλε που δημοσίως ανήγγειλε την ομοφιλοφιλία του, θα περιμέναμε μια πολύ πιο ένθερμη υποστήριξη της οδηγίας και ελπίζω τελικά να δώσει η Γερμανία την όθηση και να εγκριθεί αυτή η οδηγία. Πάντω νομίζω ότι θα πρέπει να συσπηρωθούμε όλε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, ε, γιατί τα θύματα των διακρίσεων, ε, για όποιο λόγο και αν υφίσταται τη διάκριση, θα πρέπει να δείξουν κατανόηση για τι διακρίσει και να συσπηρωθούμε σε ένα κοινό μέτωπο, που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διαιρεθεί. Δεν θα πρέπει να κάνουμε διακρίσει μεταξύ των διαφόρων ομάδων που υφίστανται διακρίσει. Σε ό,τι αφορά την ε, κοινωτική νομοθεσία κατά των καταργήσεων, πέραν της απασχόλησης, έχουμε πολλά κρατημέλη που δεν προστατεύουν ε, τους, τις λεσβίες ομοφιλόφιλους και αμφιφιλόφιλόφιλους από τις διακρίσεις. Και τέτοιες χώρες είναι η Κύπρος, η Εστονία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Πολωνία. Από τη μια άκρη της Ευρώπης μέχρι την άλλη υπάρχουν χώρες που δεν προστατεύουν ε, τους ΛΟΑ ε, Αυτέ οι κοινότητε είναι πιο ευάλωτε, υφίστανται εκφοβισμό στα σχολεία, προπυλακισμό από στρατού, από γιατρού, άρνηση παροχή περίθαλψη. μπορεί να του απαγορευτεί σε εστιατόρια ε, ή να του απαγορευτεί η διαμονή σε ξενοδοχείο μαζί με τον σύντροφο. Πολλέ φορέ θερούνται κοινωνικά επιδόματα, συντάξει. Έχω διπλή ιδιότητα γιατί είμαι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου και τη εθνική ε, Πολωνικής οργάνωση λεσβιών, ομοφιλοφίλων, φιλοφίλων και διαφιλικών που προσπαθεί να καταπολεμήσει τι διακρίσει κατά των ομοφιλοφίλων. Και εδώ και δέκα χρόνια προσπαθώ να βοηθήσω θύματα διακρίσεων και να δω πώς επιτόπου λειτουργεί αυτή η έλλειψη προστασίας. Και ένα από τα επιχειρήματα που ακούω από τις αρμόδιες πολωνικές αρχές και είναι ένα επιχείρημα που πολλοί ακτιβιστές ακούν είναι ότι οι αρχές δεν έχουν ε, τις υποθέσεις στα χέρια τους. Δηλαδή τα θύματα των διακρίσεων δεν κάνουν καταγγελίες για τις διακρίσεις που υφίστανται. Μπορώ να σας πω εκ πείρας ότι για έναν ε, νέο ομοφιλόφιλο ή μια νεαρή λεσβία φιλόφιλο ή μια νέα ριλεσβία στην ε, Πολωνία η, διάκριση είναι κάτι φυσιολογικό, είναι, είναι ένα στοιχείο της πραγματικότητας και προσπαθούν να το αντέξουν και έχουν εκπονήσει και μια στρατηγική επιβίωση. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο που φαίνεται το, το αντιμετωπίσουν σε κάτι συνηθισμένο. Έχω δει υποθέσει πρόσφατα μια νεαρή κοπέλα τη Βερόνικα που δεν αισθανόταν πολύ άνετα στην οικογένειά της στο χωριό της ήρθε στη Βαρσοβία, πήγε στη Βαρσοβία για να σπουδάσει, την πίεσαν οι γονείς της να σπουδάσει, είπαν ότι θα της πληρώσουν διαμέρισμα και όσο έμενε στη Βαρσοβία ε, βρήκε ε, μια φιλενάδα ε, και γνωρίζαμε τι θα συνέβαινε. Δεν μπόρεσε να κρύψει από τους γονείς της την ομοφιλοφιλία της. Α, της είπαν οι γονείς Ωραία, δική σου ζωή δεν πρόκειται να σου στο διαμέρισμα. Είναι 19 χρονών, μένει στη Βαρσοβία και θέλει να συζήσει με τη φίλη τη. Οπότε πρέπει να βρει ένα διαμέρισμα. Είναι φοιτήτρια όμω. Δεν έχει πολλά χρήματα, ούτε και η φίλη τη το ίδιο. Ψάχνουν λοιπόν διαμέρισμα να νοικιάσουν για να συγκατοικήσουν. Και κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά είναι ψάχνουν διαμέρισμα και ο ιδιοκτήτη όταν, ανακα... όταν ανακαλύπτει ότι η δεύτερη κοπέλα δεν είναι συγγενής, δεν είναι συμφοιτήτρια, δεν είναι φίλη, αλλά σύντροφος, αρνείται τη... το ενίκιο. Και ο ένας μετά τον άλλο οι ιδιοκτήτες της λένε δυστυχώς έχει δινικιαστεί το διαμέρισμα. Θα μπορούσε να καταγγείλει τη διάκριση αυτή στις αρχές, αλλά είναι ήδη θύμα της διάκρισης. Την έχει απορρίψει η οικογένειά της, όπως πολύ συχνά συμβαίνει ε, στην Πολωνία. Γιατί μερικές οικογένειες υποστηρίζουν τα μέλη, αλλά όχι. Δεν έχετε οικονομικά μέσα να προσφύγει στο δικαστήριο. Ήρθε σε εμά για να την στηρίξουμε. Αλλά μέχρι τα τέλη της εβδομάδα μόνη της θα πρέπει να βρει ένα δωμάτιο για να ζήσει προτιμάει να μην καταγγείλει το θέμα. Γιατί η προτεραιότητα δεν είναι να να καταγγείλει το θέμα στι αρχέ. Το... Η προτεραιότητά τη είναι να βρει ένα δωμάτιο για να μείνει. Δυστυχώ αυτά συμβαίνουν στην καθημερινότητα με τι διακρίσει. Μια άλλη ομάδα που υφίσταται πολλαπλέ διακρίσει είναι οι νεαροί ομοφυλόφιλοι. Οι διεμφυλικοί, αμφιφυλόφιλοι και λεσβείες ε, Πραγματικά ακούμε τραγικές ιστορίες στην οργάνωσή μου. Είχαμε την περίπτωση του Κούμπα που ήρθε στην Ήλγα και έγινε και εθελοντής τελικά ένα λεπτό ξανθό αγόρι που σπουδάζει ε, μαγειρική σε μια τεχνική σχολή. Μάλιστα ο δάσκαλος του ανέθεσε ως εργασία να βρει τον προπολογισμό ενός νοικοκυριού, να, να σχεδιάσει τον προπολογισμό ε, μιας ε, ε, οικογένειας με δύο παιδιά. Ο Κούμπα που είναι ομοφιλόφιλος έγραψε, σχεδίασε τον προπολογισμό για ένα νοικοκυριό στο οποίο όμως είναι δύο ομοφυλόφιλοι γονείς. Δεν το δέχτηκε αυτό ο δάσκαλος, το συζήτησε με τον Κούμπα και έφερε το θέμα στην τάξη. Λέει, φαίνεται παιδιά ότι ο Κούμπα είναι πιο έξυπνο από εσά και δεν μας έδωσε το προπολογισμό μιας οικογένεια με έναν άντρα και μια γυναίκα, αλλά με δύο γυναίκες. Τα υπόλοιπα παιδιά συμφώνησαν με τη δασκάλα και συνέχισαν να παρενοχλούν και να εκφοβίζουν τον Κούμπα. Ο Κούμπα παραπονέθηκε στο διευθυντή, και ο διευθύντη είπε στο σχολείο μα: κανένας ε, δεν έχει υποστεί ξυλοδαρμό, κανένας δεν έχει υποστεί εκφοβισμό. Φαίνεται βλέπει πολλέ αμερικανικέ ταινίε για τέτοια ομοφοβική συμπεριφορά. Αυτό είπε λοιπόν ο διευθυντής του σχολείου. Αλλά και το Συμβούλιο Γονέων είπε τι να, ο ψυχολόγο είπε τι να σου πω. Δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτή την αντίσταση στα σχολεία. Το μόνο είναι να σε βοηθήσει να γίνει λίγο πιο σκληρό, να αντέχει καλύτερα αυτό τον εκφοβισμό εκπρόσωπος ε, των ε, δικαιωμάτων των ε, φοιτητών, ο διαμεσολαβητής κατά κάποιο τρόπο, συνήγορος του φοιτητή, του μαθητή, είπε στον Κούβα «Εσύ φταίς, δεν πρέπει να διατυμπανίζεις και την ομοφιλοφιλία σου». Αυτή είναι η περίπτωση λοιπόν του Κούμπα Μπορεί ο Κούμπα να έρθει στην οργάνωση να καταγγείλει το θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά εδώ μιλούμε ουσιαστικά για δύο εφήβους που αντιμετωπίζουν ε, τέτοιες διακρίσεις στο πετσί τους καθημερινά. Για πολλά χρόνια η Πολωνία ήταν από τις πιο ομόφοβες ε, χώρες στην, στην Ευρώπη και παρακολούθησε πολλές δημόσιες ακροάσεις στην Ευρώπη και από όλη την Ευρώπη αναφερόταν η Ισπανία ως καλό παράδειγμα και η Πολωνία ως ε, αρνητικό παράδειγμα. μία χώρα παράδεισος και άλλη ως κόλαση για τους ομοφιλόφιλους. Κάναμε λοιπόν, ε, ασκήσαμε πιέσεις, ε, κάναμε lobbying και συνεργαστήκαμε και με άλλες οργανώσεις ισότητας στην Πολωνία και καταφέραμε να περάσει ένα νομοσχέδιο κατά των διακρίσεων στην Πολωνία. Βέβαια δεν είχαμε ούτε έχουμε μια οριζόντια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάναμε λοιπόν ε, ε, τοπικά τις προσπάθειές μας και ασκήσαμε πιέσεις ε, για να προοδεύσει η Πολωνία. Από το 2005-2006 πολλά έχουν αλλάξει, πολύ πρόοδο έχει σημειώσει η πατρίδα μου και το 2011 σας τύπωσε εδώ μία νομοθετική πράξη που ενσωματώνει κάποιες από τις κοινοτικές διατάξεις ίσης μεταχείρισης. Ο αρμόδιος Υπουργός Ισότητας είπε όντως υπάρχουν κάποιες κοινοτικές οδηγίες που καλό θα είναι να εφαρμόσουμε και ειδού τη λάβαμε 10 σελίδες ε, με την πολωνική νομοθετική πράξη που εφαρμόζει κάποιες κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις. 10 σελίδες. Τις διάβασα το πρωί και ε, σημείωσα με μαρκαδόρο ποιες εξασφαλίζουν προστασία για τους ομοφιλόφιλους, λεσβίες, αμφιφιλοφιλόφιλους. Βλέπετε, το τόνισα με πορτοκαλί μαρκαδόρο. Ε, περίμενα, περίμενα λοιπόν, ξεράθηκε ο μαρκαδόρος και γιατί δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Μόνο σε περίπτωση επασχόλησης προστατεύονται ουσιαστικά οι ΛΟΑ. Τίποτα δηλαδή, καμία προστασία ουσιαστικά. Ελάχιστη διαφορά για τις διακρίσεις ε, κατά των ομοφιλοφίλων. Η χώρα μου είναι μία από τις χώρες που δυστυχώς ε, δεν έχουν ε, προστασία κατά των διακρίσεων λόγω ε, γενετήσιου προσανατολισμού. Και χώρες που δεν έχουν τέτοια νομοθεσία δεν πρόκειται από μόνες τους να αναλάβουν την πρωτοβουλία για να τη θεσπίσουν. Ό,τι και να κάνουμε εμείς τοπικά ε, με λόμπι, με πιέσεις, δεν πρόκειται να τελεσφορήσει αν δεν έχουμε μία ε, πανευρωπαϊκή, κοινοτική, δεσμευτική οδηγία που είναι υποχρόνη τις ε, απρόθυμες χώρες να θετήσουν τέτοιες ε, διατάξεις κατά των διακρίσεων. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει το σήμα στα κράτη-μέλη ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια οδηγία, ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια τέτοια οδηγία και να υπάρξει και τεχνική υποστήριξη της ομάδας εργασίας για τα κοινωνικά ζητήματα. Να δούμε για παράδειγμα ε, μια σύγκριση μεταξύ του κόστους ε, της διάκρισης και του κόστους της εφαρμογής της οδηγίας. Συμφωνώ με τον κύριο Μπορό ότι δεν θα πρέπει η συζήτηση να παρεκτραπεί σε οικονομικά θέματα. Δεν είναι συζήτηση μόνο για τα λεφτά, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό επιχείρημα για να πείσουμε τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη, να έχουν διαβουλεύσει με μη κυβερνητικέ οργανώσεις πριν τι συνεδριάσει στην ομάδα εργασία και στη συνεργασία με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα πρέπει να φροντίσουν να μην ε, ε, αλλοιώσουν το κείμενο και να μην αφαιρέσουν κάποιους λόγους διακρίσεων, κάνοντας το πιο ασθενές. Επίσης, η συμμαχία των πιο προοδευτικών χωρών που είναι υπέρ της οδηγίας θα πρέπει να πιέσουν πιο έντονα για να εγκριθεί η οδηγία αυτή και από τις υπόλοιπες πιο διστακτικές χώρες αλλά και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση να συνεχίσουν να, βο... να βολιδοσκοπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πιέζουν με ερωτήσει και να προωθούν την οδηγία. Όπως είπα, η Πολωνία για πάρα πολύ καιρό ήταν ένα σκοτεινό σημείο σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις κατά τον ΛΟΑΔ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Είμαι αρκετά αισιόδοξο και ελπίζω όλοι οι θύνοντες να μου υποσχεθούν ότι μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια θα έχουμε διεκπαιρεώσει την έγκριση οδηγία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά και ας ολοκληρώσουμε αυτόν τον γύρο με, τις, ε, με τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν ε, τον γύρο με τον τέταρτο ομιλητή για τη, ε, για τη θρησκεία, ο κύριος ε, Μιχαήλ Πριβό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω τη χαρά σήμερα να εκπροσωπώ την οργάνωσή μου που αντιπροσωπεύει πάνω από 700 οργανώσεις στην Ένωση που καταπολεμούν τις διακρίσεις με βάση την εθνότητα και την αλλά και τις ε, θρησκευτικέ μειονότητες. Ε, είδαμε ότι όταν πρόκειται για μειονότητες αυτά τα θέματα αλληλοκαλύπτονται. Όπω είπε η συνάδελφο Σοπέν σήμερα το πρωί, η ΕΝΑΡ, η οργάνωσή μου, ιδρύθηκε από ένα μεγάλο αριθμό οργανώσεων που είχαν αποτελέσει το Standing Line Group. Είχαμε λοιπόν στις μνήμες μας ε, αυτόν τον αγώνα για την ισότητα με βάση το άρθρο 13 της Συνθήκης και τις οδηγίες για την ε, ισότητα στην εργασία και, στην, ε, και την ισότητα στους, σε φορά την φυλή. Θέλησαμε λοιπόν να υπάρξει ένα πακέτο, αλλά δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί και σήμερα η χολή, θα έλεγα, ε, νομοθεσία που έχουμε οφείλεται σε αυτή ακριβώς την ε, έλλειψη επιθυμίας ε, όλων των κρατών μελών που θα θέλουν να καλύψουν πολλά θέματα, π.χ. ομοφιλοφιλία και θρησκεία. Ακούστηκαν λοιπόν πολλές λεπτομέρειες σήμερα, πολλές προφορίες για τεχνικά θεσμήματα, τα οποία ε, συζητήθηκαν στο πλαίσιο των οδηγιών. Δεν θα μιλήσω τεχνικά, ε, αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας, αλλά και θα ήθελα το χρόνο που έχω στη διάθεσή μας να κάνω μια ανάγνωση πολιτικής φύσης ε, και διότι έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει κάτι το παράλογο για την μη έγκριση της οδηγίας. Τα επιχειρήματα υπάρχουν εδώ, υπάρχουν επιτόπιτο, δεν πούμε παραπάνω, αλλά και όμως ε, υπάρχει εμπλοκή από το, εδώ και 15 χρόνια, θα μπορούμε να βρεθούμε στο 1997, μας ε, ε, μιλούν για διάφορα προβλήματα. Τότε ήταν το ζήτημα των σχολείων, τη θρησκεία, των οργανώσεων για τη συμπερίληψη ε, προσώπων με διαφορετική θρησκεία ή με διαφορετικό γεννήσιο προσανατολισμό σήμερα είναι το θέμα τη αναπηρία που μα απασχολεί. Είναι παράδοξο, το θυμόμαστε το 2007 ο πρόεδρο Μπαρόζο είχε προτείνει ε, αισθανόμενο στην εμπλοκή να μην προχωρήσει, να προχωρήσει με μια οδηγία που θα καλύπτει μόνο την αναπηρία. Γιατί το 2007 θα μπορούσε να γίνει, να, γίνει, να συμβεί κάτι και σήμερα δεν είναι πλέον δυνατόν. Ακούμε διάφορους απόϊχους, ε, βυζαντινές βυζαντινολογίες στο Συμβούλιο σχετικά με την προσβασιμότητα για το θέμα της ε, οικολογικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει ε, τη χρήση ε, άμμου κλπ. Όλα αυτά πραγματικά είναι μπουρδες, συγγνώμη που το λέω. και επίσης αναφέρεται και η επιπλέον εις βάρος των αναπήρων ανθρώπων αυτών που, που αισθάνονται τον οικονομικό τον πολιτικό αποκλεισμό και τους δίνουμε να καταλάβουν ότι είναι και κόστος στην κοινωνία μας και τώρα έχουμε και την χειροπέδη για τον πρόοδο των δικαιωμάτων των υπολείπων. Θέλω λοιπόν ότι είναι εύκολο σήμερα να παραμείνουμε κλεισμένοι σε έναν υπολογισμό ε, καθαρά λογιστικό πόσο κοστίζει άχι εκατομμύρια Δυστυχώ δεν μπορούμε διότι δεν υπάρχουν χρήματα κρίση κλπ μας κοροϊδεύουν δεν είναι αυτός ο λόγος ε, όπως είπε και ο συνάδελφός μου σήμερα το πρωί είναι πως η ισότητα αφορά όλους 100% είμαστε νέοι γυράσκουμε. Σήμερα έχουμε καλή υγεία. Σε μια δεύτερη φάση μπορεί να γίνω ανάπηρο. Μπορώ, να, αλλάξω φύλλο, μπορώ να αλλάξω θρησκεία, μπορώ να αλλάξω ακόμα και χρώμα, της ε, σάρκας μου. Είμαστε πλούσιοι σήμερα, φτωχοί αύριο. Στην ουσία το ζήτημα της ισότητας ε, ως ενεργό προστασία των ε, πλέον αδυνάμων της κοινωνίας μας επιφέρει και το ζήτημα της αναθεώρησης της ιδέας περί ανακατανομής του πλούτου αλλά και την παροχή ενός αυξημένου αριθμού κοινωνικών υπηρεσιών. Εδώ έγκυται το πρόβλημα για, για μας. Οι κοινωνίε μας δεν ήταν ποτέ τόσο πλούσιες όσο σήμερα. Αν δούμε την πρόοδο του γαλλικού ΑΕΠ σε σχέση με το 2010, σήμερα βρισκόμαστε 2-3 εκατομμύρια 800 δολάρια με πρόοδο 10%. Στη Γερμανία έχει το αυξήσει το ΑΕΠ τους 10% ε, σε σχέση με το 2010. Πού είναι η κρίση ή τουλάχιστον για ποιον είναι κρίση. Αυτό το οποίο είναι προβληματικό είναι η κατανομή των ε, ωφελών ε, σε αυτή την κοινωνία. Και όσοι αντιτίθεται στην οδηγία και όσοι αρχίζουν να μιλάνε για θέματα επικουρικότητας κλπ. καταλαβαίνουμε πολύ καλά ε, γιατί το κάνουν. Όταν μιλάμε για δέκα δις, ε, στην ουσία είναι ε, μια λεπτομέρεια. Εάν η προσέγγιση, όπως είπε ο Ραούλ Ρεμέβα σήμερα, είναι η υλοποίηση μιας ε, κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, που επιθυμεί να υλοποιούνται όλα τα δικαιώματα υπέρ των πολιτών, στην Ευρώπη έχουν του καλύτερου νομομαθείς, μπορούν να βρουν τι καλύτερε διατυπώσεις. Και όταν επανερχόμαστε στο θέμα του κόστου που συνδέεται με ζητήματα ισότητα και όχι μόνο σε αφορά την προτασιμότητα για τους αναπήρους, θα πρέπει να δούμε ότι πρόκειται μόνο για δημόσιες επενδύσεις που συμμετέχουν στην ΕΦΗ και χωρίς αποκλεισμούς ε, Ευρώπη 2020. Αυτές λοιπόν οι επενδύσεις ε, στην ουσία είναι εξίσου σημαντικές με τα χρήματα τα οποία χορηγούμε στην ΚΑΠ και κανείς δεν αφισβητεί τόσο καλές όσο αυτά τα οποία δαπανούμε στην ενέργειες ενέργειας ε, ακόμα και με τα δισεκατομμύρια ευρώ που παρέχονται σε επιχειρήσεις άμεσα ή έμεσα μέσω των επιδοτούμενων ε, ε, θέσεων εργασίας. Όλοι οι επενδυτές εποφελούν από αυτό. Στην Ευρώπη, ε, η εμεσα μεσω των επιδοτουμενων θεσεων εργασία. ολοι οι επενδυτες εποφελουν απο αυτο η οικονομια επιδοτείται από τον δημόσιο. Γιατί λοιπόν μας δημιουργούν πρόβλημα όταν ζητάμε μερικά δισεκατομμύρια για λόγους προασιμότητας. Υπάρχουν λύσεις λοιπόν. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις το έχουν αποδείξει αλλά επανερχόμαστε πάντα στο ζήτημα της πολιτικής βούλησης. Θέλουν ναι ή όχι μια Ευρώπη δίχως αποκλεισμού όπου όλοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και θα μπορούν να οδηγηθούν σε ανάταση πνευματική και όχι μόνο. Λοιπόν, κλείνοντας να πω ότι όλες οι συζητήσεις ε, που είχαμε τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμεύουν παρά να ε, διασκεδάζουν ε, τις ε, ανησυχίες κάποιων και να προστατεύουν τα συμφέροντα όσων πιστεύουν ότι η ισότητα στην ουσία είναι κακή για τις business, δεν επιτρέπει την εκμετάλλευση και ιδίως δεν επιτρέπει πολύ υψηλά ποσοστά κέρδους εμείς εδώ σήμερα για όλους όσους προσωπούμε οι οποίοι ψοφάνε στον δρόμο, συγγνώμη για την έκφραση, εν τη σιωπή ενώπιον αυτής της ε, στάσης ε, τόσο κάποιων κρατομελών, ε, κάποιων τμήματων της Κομισιόν, αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί ακούσαμε κάποιες φωνές που δεν εκφράστηκαν απόλυτα υπέρ, αν και το Κοινοβούλιο στο σύνολό του είναι υπέρ και το μήνυμά μας είναι σαφές. Θα πρέπει να διαλέξουμε τον το δρόμο μας, συγγνώμη, δεν ε, θέλω να είμαι μανιχαϊστής, αλλά σε ό,τι φορά ισότητα δεν υπάρχει μέση οδός. Είμαστε υπέρ, είμαστε κατά. Δεν υπάρχει κάτι τον διάμεσο. Θα πούμε σήμερα ότι οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι, όποια και είναι ο θεσμός των οποίων ανήκουν, θα πρέπει να επιλέξουν ε, ή την ε, ισότητα και πρόοδο για όλους ή την, την διακρίσεις και αυτό το οποίο τελικά θα αποβεί ε, προ όφελο ορισμένου και όχι του συνόλου. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ και όλου του υπόλοιπου προσκεκλημένου. Ε, ολοκλώσαμε τι παρουσιάσει. Έχουμε μερικά... Λίγα λεπτά ακόμα για έναν ε, τρίτο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιος ευρωβουλευτής που να θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Κλέης, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ συγκεκριμένα να θέσω ένα ερώτημα προς τον κύριο Ντεβίτε. Πριν ε, κάποιες εβδομάδες ε, νομίζω αναφέρθηκε στις ειδήσει. Είχε γίνει προσφυγή κατά της ε, οργάνωσής του, της Equinet. Σε ένα μεγάλο ε, Ολλανδικό πολυκατάστημα. Υπήρχε πρόβλημα με μια εργαζομένη που εμφανίστηκε με μαντίλα και αρνήθηκε να τη βγάλει παρότι είχαν παραπονεθεί ε, πελάτες και τελικά απολύθηκε. Η χέμα ήταν ε, η επιχείρηση. Δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα διάκρισης για θρησκευτικούς λόγους. Απλά όλοι οι υπάλληλοι έπρεπε να είναι απολύτως ε, ουδέτεροι όταν εργάζονταν στο κατάστημα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η θέση του κύριου Ντεβίτε, ε, διότι όχι... Ε, μόνο προσέφυγε, αλλά ε, υπήρχε και γνωμοδότηση να γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, για να υπάρξει νομολογία, δηλαδή να αλλάξει η νομοθεσία. Ένας εργαζόμενος Ε, μπορεί να αναμένεται ότι θα περιορίσει στον ιδιωτικό του χώρο τα ε, θρησκευτικά σύμβολα της ε, μπορεί να κάνει θρησκευτικέ δηλώσεις απέναντι σε συναδέρφους ή σε πελάτες. Νομίζω ότι ο κύριος Ντεβίτα έχει σαφές, σαφείς απόψεις για το θέμα αυτό. Είναι σαφής η θέση που παίρνει. Άλλωστε οι φορολογούμενοι πληρώνουν για την οργάνωσή του, διότι ε, λαμβάνει χρήματα από την κυβέρνηση. Το να ε, φέρνουμε στη, σε ακραία σημεία την ε, πολιτική ορθότητα, ε, μήπως υπονομεύει τα θέματα διακρίσεων και η οργάνωση για την οποία μιλάμε δεν υποκαθιστά τον νομοθέτη. αποφασίζοντας να φτιάξει δικούς της νόμους. Στον προηγούμενο γύρο μιλήσαμε για την αντίθεση κρατών μελών στην ε, υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας ε, κατά των διακρίσεων. Αλλά τέτοιες περιπτώσεις συμβάλλουν στις ανησυχίες των κρατών μελών. Ε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι πολύ ε, αόριστη όσον αφορά τις ε, αντιρρήσεις των κρατών μελών. Η φερόμενη αυτή ε, ε αντίθεση στο, στην, στους κανόνες είναι λίγο ε, αμφίβολη διότι ε, δεν την ε, απέλησαν για θρησκευτικούς λόγους, απλά έπρεπε, ήθελε εκείνη οπωσδήποτε να φορέσει τη μαντήλα παρά τους κανόνες σε μια τέτοια περίπτωση δεν νομίζω ότι πρέπει κανεί με τέτοιο τρόπο να εκφράζει πολιτικέ θρησκευτικέ θέσει. Προτού να δώσω το λόγο στον κύριο Ντεβίτ για να απαντήσει ή να ε, ολοκληρώσουμε τι ερωτήσει. Κυρία Κιόνι, θέλετε το λόγο. ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση προ τη Δανέζικη Προεδρία. Ε, δεν ήμουν εδώ στην αρχή τη συζήτηση. Θα ήθελα όμω από τη Δανέζικη Προεδρία να ακούσω ποιες πιστεύουν ότι είναι οι πιθανότητες να προχωρήσουμε και να ξεμπλοκάρει η ε, οδηγία κατά των ε, διακρίσεων στο Συμβούλιο. Είμαι η μόνη ε, σοσιαλδημοκράτησα στο, στην αίθουσα. Και εγώ λέει ο πρόεδρος. Ναι, αλλά ο πρόεδρος πρέπει να είναι ουδέτερος, λέει ο Μιλήτρια. Αλλά σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Θα ήθελα πολύ να ακούσω από την Δανέζικη Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σορομέβα, παρακαλώ. Θέλετε να κάνετε μια ερώτηση. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη προς την Equinet. Ε, είχατε περικοπές στον προϋπολογισμό ε, λόγω της παρούσας κατάστασης και ποιος είναι ο αντίκτυπος εάν ε, έχουν γίνει περικοπές και επίσης ε, προς το Συμβούλιο μια ερώτηση-πρόταση προ την Δανέζικη Προεδρία. Αν συμφωνούμε όλοι ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό, πιστεύετε ότι μία ή δύο συναντήσεις στο εξάμεινο αρκούν. Αν εμείς θέλουμε τόσο πολύ να προχωρήσουμε, Μήπως θα ήταν δυνατόν ή μήπως θα ήταν σοφότερο να συναντιόμαστε πιο συχνά και όπως είπανε πολλές από τις οργανώσεις ε, να ακούμε εμπειρογνώμονες σε διάφορα θέματα. Για να εμπαθύνουμε περισσότερο στο θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο. να δώσουμε το λόγο πρώτα στον κύριο Ντεβίτε, με αντίστροφη σειρά, κατόπιν στην ε, Δανέζικη Προεδρία θα δώσουμε το λόγο και ε, στο Συμβούλιο τέτοια ερώτηση. Ο κύριος Ντεβίτε. Ευχαριστώ. Μια και η ερώτηση επιβλήθη στα Ολλανδικά, θα απαντήσω και εγώ Ολλανδικά. Καταρχήν, κάποια σχόλια. Γιατί αναφερθήκατε στη θέση μας Προέδρου της Εκουινέτ. Δεν νομίζω ότι ε, είναι σκόπιμο να έχουμε μια εσωτερική βελγική συζήτηση. Επίσης αναφερθήκατε ε, στη σχέση εργοδότη και εργαζόμενου. Αλλά εδώ ε, μιλάμε περισσότερο για αγαθά και υπηρεσίες. Αν εν πάση περιπτώσει, αναφερθώ σε ορισμένα σκέλη της ερώτησής σας. Είπατε ότι θέλουμε να τροποποιήσουμε την νομοθεσία. Πώς μια προσφυγή στο δικαστήριο μπορεί να εξομοιωθεί με προσπάθεια τροποποίηση της νομοθεσίας. Εφόσον υπάρχει νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί και αρμόδιος να επιβάλλει να φροντίσει για την εφαρμογή μιας νομοθεσίας είναι ο δικαστής σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επανέρχομαι τώρα σε αυτό που είπατε για το... Φορούσε μαντήλα υπάλληλο. Ελπίζω ε, ότι εσείς και το, σώμα, το, το κόμμα σας που κόπτεστε για την ελευθερία και την ελευθερία έκφρασης να είστε ανοιχτοί και προοδευτικοί και σε θρησκευτικά ζητήματα. Και σίγουρα η ανεξιθρησκεία θα πρέπει να ε, επικρατήσει και να μην περιοριστεί η ελευθερία θρησκείας ε, μόνο στους στίχους μιας κατοικίας. Δεν το αντιλαμβάνεται έτσι ούτε η σύμβαση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε ο σχετικός χάρτης των Ηνωμένων ε, των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ούτε στην Ολλανδία είναι ουδέτερες οι χώρες, ούτε προσπαθούν ε, στο Βέλγιο να είναι ουδέτερες. Τι γίνεται με την οικία, την Κρόιτβατ, οι άλλες ε, εταιρείε που δεν επιμένουν τόσο πολύ στη Μαντή, δηλαδή την κάνουν λάβαρο. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά πού το πάτε. Έχουμε μία εντολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγξουμε τέτοιες υποθέσεις και νομίζω ότι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και ανταπεξερχόμαστε στις υποχρεώσεις μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πολλοί φορείς ισότητας, κύριε Ρωμέβα Ερόεδα, υπέστησαν τις αρνητικές συνέπειε των δημοσιονομικών περικοπών. Αυτό είναι φυσικά αναπόφευκτο σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Εμεί δεν πιστεύουμε ότι η λιγότερη ισότητα είναι η απάντηση ε, στην οικονομική κρίση. Γιατί οι μελέτες δείχνουν ότι η αύξηση του ΑΕΠ ε, κατά 15% θα γίνει δυνατή ε, και μόνο και με την εφαρμογή της ισότητας. Ποιο μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ε, με την εφαρμογή αυτών των μέτρων θα έχουμε 15% αύξηση του ΑΕΠ και ότι η πρόθεση της ισότητας θα εξυπηρετήσει και την οικονομία και θα οδηγήσει σε άνθηση κατά καθάκια της τις Ωραία, σας ευχαριστώ. Ίσως κάποιος από το Συμβούλιο, εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας, θα ήθελε να απαντήσει στην ερώτηση που τέθηκε για το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ρωτήσατε ποιες είναι οι προβλέψεις μας για την πρόοδο των εργασιών στην οδηγία αυτή στη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας. Μακάρι να μπορούσα να σας απαντήσω με αισιοδοξία και πολύ φιλοδοξία, αλλά επειδή είμαι και ρεαλίστρια, δεν έχω και μεγάλες ελπίδες. Βλέπουμε την πορεία της οδηγίας την τελευταία τετραετία και δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Πόρο απέχουμε από τη διεκπαιρέωση των εργασιών. Όπως είπαμε και προηγουμένως και τεχνικές εκκρεμότητες υπάρχουν και πολιτικά προβλήματα. Ε, αν θα απαντούσα και στον εισηγητή ότι στο ερώτημα αρκούν δύο συζητήσεις, δύο συναντήσεις το εξάμεινο. Φυσικά και δεν αρκούν. Και πέραν των νομικών επιπτώσεων και των δημοσιονομικών επιπτώσεων και της αντίδρασης ε, ή της ε, αντίθεσης ορισμένων χωρών, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα το θέμα αυτό δεν είναι υψηλή προτεραιότητα πια για πολλέ χώρε μέλη. Χάθηκε η ορμή που υπήρχε προηγουμένω. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πάντω αυτή είναι η αίσθηση ότι έχει χαθεί η ορμή που είχαμε προηγουμένω. Και αυτό ήταν πρόβλημα και για μας όταν διαλέξαμε τις προτεραιότητες της Δανικής Προεδρίας. Προσπαθήσαμε να σφιγομετρήσουμε και τα κράτη-μέλη για να δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε την αίσθηση ότι είναι μεγάλο πρόβλημα σαν τιτανικό σε αυτό το θέμα. Προς το παρόν αυτό το χαρακτήρα έχει και δεν μπορούμε μόνοι μας να πλοηγήσουμε ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα. Θα χρειαστούμε την υποστήριξη ε, των χωρών μελών. Υπάρχουν χώρες που είναι υπέρ, αλλά επαναλαμβάνω δεν υπάρχει αυτή η όθηση. Είναι η ατμόσφαιρα που επικρατεί προς το τέλος της γιορτής, όπου όλοι είναι κάπως κουρασμένοι και δεν ξέρουν, δεν έχουν πια την, τη ζέση και την, τον ενθουσιασμό που είχαν στην αρχή. Αυτή την αίσθηση έχουμε κι εμείς για την πορεία αυτών των συζητήσεων. Πιστεύω ότι πόρο απέχουμε από την ανέβρεση λύσης. Κύριε Πριβό, θέλετε να δώσετε μια απάντηση στα ζητήματα θρησκευτικών διακρίσεων που έθεσε ο κύριος Κλέης. Δεν πρόκειται για απάντηση, ερώτηση. Ήσασταν ε, πολύ απόλυτος ε, στο ότι αυτός ο υπάλληλο ε, έδινε την εντύπωση ότι δεν ήταν ουδέτερος τώρα κατά τα υπόλοιπα συμφωνώ με τον κύριο Ντεοβίτ αλλά θα ήθελα να γνωρίζω και μπορούμε να το συζητήσουμε και εκτός ε, ενώπιση Αλλά αφορά το ζήτημα των διαθροτικών διακρίσεων που μας απασχολούν. Πού, σε ποιο benchmark, σε ποιο σημείο αναφορά ε, αναφέρεστε όταν λέτε ότι η στάση είναι ουδέτερη. Αν έχετε κάποιους δείκτες ε, θα ήθελα να τους ακούσω. Θα βοηθούσε στη συζήτηση κύριε Κλάης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε εγώ δεν εκπροσωπώ την ΕΜΑ και άρα μπορώ να απαντήσω γιατί στο κατοχώρης κάτι γίνεται και στη Φιλανδρά όχι, το αντίστροφο. Θεωρώ ότι είναι καλό που έχει αυτό το δικαίωμα ελεύθερης ε, άποψης. Δεν ήταν ε, πάντα κάτι που ίσχυε στην οργάνωσή σας. Ε, σκέφτομαι για κάποιες δικαστικές διαδικασίες που αναλάβατε και κατά πολιτικών κομμάτων και ιδιαίτερα κατά του δικού μου. Με στους τα ξέρετε πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Τώρα η συζήτηση δεν αφορά αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι να γνωρίζουμε κατά πόσον ένας υπάλληλο, ένας ε, εργοδότης μπορεί να ζητήσει από το προσωπικό του να κατά την ώρα παρουσίας του στο χώρο εργασίας να μην ε, ε, ασκούν πολιτική είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εργασία που τους έχει ανατεθεί. Δηλαδή εγώ, παράδειγμα, όταν είμαι σε επαφή με πελάτες ε, σε μια επιχείρηση, να προσπαθήσω να διαφημίσω το κόμμα μου, να, προσπαθήσω, να τους προσιλητήσω σε ένα κόμμα ή σε ένα κίνημα το οποίο συμμετέχω. Νομίζω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει στον χώρο εργασίας. Είναι κάτι που πρέπει να γίνεται εκτός επιχείρησης. Η επιχείρηση πρέπει να είναι ουδέτερη απέναντι στους πελάτες προκειμένου να μην δημιουργούνται πολεμικές ε, παρανοήσεις, παρεξηγήσεις κλπ. Για να συμβεί λοιπόν αυτό θα πρέπει στο χώρο εργασία να είμαστε ουδέτεροι. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η διαφορετικότητα γίνεται αποδεκτή, μπορεί να οδηγήσει φυσικά σε ε, αντιπαραθέσεις ε, και συγκρούσεις, ε, αλλά ο εργοδότης μπορεί και να απαιτήσει από το προσωπικό του να μην ασχολείται με την πολιτική κατά τον χρόνο εργασίας. Ξέρετε πολύ καλά, όπως και εγώ, ότι οι δικαστές χάρη στην ερμηνεία που δίνουν σε ένα νομοθετικό κείμενο μπορούν να θέσουν κάποια, μια περίμετρο, κάποια, όρια, αν το εύρος το εύρο εφαρμογή, το πεδίο εφαρμογή Ναι, μπορούν να το επεκτείνουν ή και να το περιορίσουν. Χάρη λοιπόν σε αυτό το περιθώριο ερμηνείας που έχουν. Και αν ένα προδικαστικό ζήτημα υποβάλλεται, λαμβάνεται μια απόφαση, ένα βούλευμα, το οποίο όμως και αυτό μπορεί να ερμηνευθεί με τρόπο διαφορετικό. Υπάρχει μια νομολογία περί αυτού. Ε, διότι δημιουργούμε προηγούμενα. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο εσείς παρεμβαίνετε. Διότι οι προσφυγές που θα γίνουν μετά από την απόφαση θα ε, συμπεριληφθούν ε, στην νομολογία και κινδυνεύουμε να έχουμε εδώ μια κυβέρνηση δικαστών. Εάν τους αφήσουμε απόλυτη ελευθερία μπορούμε να θέσουμε στο στο δικαστήριο του Στρασβούρου τα για ανθρώπινα δικαιώματα και μπορούμε να έχουμε μια εφαρμογή πολύ περιοριστική της, της, πολιτικής, πολιτικής. Και, ναι, κοιτάξτε, εδώ είμαστε κοινοβουλευτικό όργανο και κάθε μέλος του κοινοβουλίου έχει το δικαίωμα να εκφράζεται, να εκφράζει τι απόψει του και δεν ε, μπορούμε να τι αμφισβητήσουμε τώρα. Εάν εσεί θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο ως προσκεκλημένο σε αυτή την ακρόαση, Σα καλώ να το πράξετε, αλλά ήθελα να σας ζητήσω να μην ε, αρχίσετε μία συζήτηση, μία αντιπαράθεση σε αυτήν την φάση της ακρόασης. Ευχαριστώ Πρόεδρε πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι αυτό ήταν ένα βαριικό ερώτημα. Θα ήθελα ως εκ τούτου να ζητήσω από τον κύριο Κλάις να συζητήσουμε εντάξει και να του δώσω κάποιες απαντήσεις. Δεν θέλω λοιπόν να μπω σε μια συζήτηση. Αλλά όταν μιλάμε για αγαθά και υπηρεσίες, τι εννοούμε ουδέτερο σε ένα εστιατόριο. Τι σημαίνει ουδέτερο στο ε, δημόσιες μεταφορές και τι σημαίνει να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους ε, ουδέτερα όταν πρόκειται για προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να γύρουμε. Έχουμε ένα ε, εστιατόριο, μπορούμε να ζητήσουμε, να απαγορεύσουμε μάλλον στους πελάτες να, να είναι ομοφιλόφιλοι παρατήρηση εκτός μικροφώνου. Ωραία. Σας ευχαριστώ κύριε Ντεβίτε και φυσικά σας ε, ευχαριστούμε για τον τρόπο με τον οποίο ε, συμμετείχα στη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους, ε, αλλά πρωτού να περάσουμε στα τελικές, τελικά σχόλια που θα τα κάνει ο κύριος εισηγητής λάβαμε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον κύριο Ολιβιέντε Σούτερ ο οποίος είχε προσκληθεί στη σημερινή ακρόαση δεν τα κατάφερε όμως όπως σας είπα αλλά θέλει να μας ότι κάποια στοιχεία της ε, παρουσίασης που θα ήθελα να κάνει η οποία θα διαρκούσε 15 λεπτά και να σας πω ότι είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ της Επιτροπής μας δηλαδή και επιθυμεί να σας πω ότι θεωρεί ότι ένα εναρμονισμένο επίπεδο προστασία ε, σε θέματα διακρίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης ε, θα αποτελούσε σημαντικό πλεονέκτημα όπως εναρμόνιση μετά από την πρόταση για οριζόντια οδηγία που έγινε από την Κομισιόν την άρση των διακρίσεων των άμεσων και των έμεσων που δεν αφορούν ε, την ιδιωτική ζωή και αυτό θα ήταν συνεπές ε, με τα κοινωνικά δικαιώματα, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, την νομολογία του, νομοθεσία του Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα διευκολύνει την άσκηση των ε, δικαιωμάτων και παράλληλα την ε, ελεύθερη πρόσβαση αγαθών ε, μεταφορών, εκπαίδευση κλπ. Και ο καλύτερος τρόπος για να συμβάλλουμε, σύμφωνα με την παρουσίαση του κ. Ολβιέντε Σούντερ, θα ήταν να μελετήσουμε τη σύνδεση μεταξύ πρόσβασης ε, στην αγορά και την ε, προϊόντων ε, εργασία, στην εργασία, πρόσβαση σε άλλα αγαθά που αναφέρονται στο άρθρο 3 And the racial equality και την οδηγία περισσότητας για την επιδευξή πραγματικών ίσων ευκαιριών. Λυπάται λοιπόν που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα ανάμεσά μας και είναι στη διάθεση όλων των μερών της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ διοδήποτε τρόπου. Λοιπόν, ακούσαμε αυτά που, μας, ε, που ήθελε μάλλον να μας πει ο κύριος Ντεσούτερ. Ακούσουμε τώρα και τα συμπεράσματα του εισηγητή κύριου Ρωμένα. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, διότι σχεδόν όλα υπόθηκαν. Απλά, εν είδη σύνοψης, καταρχήν θα ήθελα να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω ε, τους, όλους, όλους τους ομιλητές για τη συμβολή τους, διότι όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα είναι πράγματα που πρέπει να υποθούν. Και αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα που θα ήθελα να εξάγω. Ο βασικός λόγος που κάνουμε εμείς αυτή την ακρόαση είναι τα απόλυτα σαφή στοιχεία που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή που δείχνουν ότι η έλλειψη μιας τέτοιας οδηγίας ε, δημιουργεί δυσκολίες στη ζωή πολλών ε, πολιτών μας, ε, φίλων, συναδέρφων, ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά. Υπάρχουν σαφή στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό είναι κάτι απαραίτητο. Δεύτερον, χρήσιμο ήταν για μένα, χρήσιμη ήταν για μένα η επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα για την υιοθέτηση αυτής της οδηγίας, μάλλον το αντίθετο. Υπάρχει νομική ανάγκη να έχουμε αυτό το νομοθέτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εφαρμοστεί. Η μη ύπαρξη αυτής της οδηγίας, κατά τη γνώμη μου, αντίκειται στη, στη βάση της ε, συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ελεύθερη κινητικότητα και άλλα δικαιώματα. Για μένα αυτό είναι σαφές. Υπάρχει λοιπόν νομική ανάγκη και πολλά στοιχεία που μας το δείχνουν αυτό. Και τέλος ε, καταλήγουμε στο πρόβλημα το οποίο είναι η πολιτική βούληση. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Από ό,τι κατάλαβα, ως κοινοβούλιο και ως κοινωνία των πολιτών, δηλαδή και οι μη οργανώσεις, μπορούμε όλοι να επικεντρωθούμε στις κυβερνήσεις ε, που ε, χρησιμοποιούν επιχειρήματα για να αντισταθούν στην οδηγία αυτό, αυτή. Θα αναφέρω τις χώρες αυτές. Ε, ε, ήδη αναφέρθηκαν η Γερμανία για λόγους κόστους, η Λιθουανία, η Τσεχία όσον αφορά τα άτομα ΛΟΑΔ. Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι πολίτες των χωρών τους αναγνωρίζουν ότι ο λόγος που δεν μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν στη Γερμανία είναι ότι η κυβέρνησή τους αντίκειται ε, στο να υπάρξει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικό είναι λοιπόν να διαδοθούν όλα αυτά τα στοιχεία ε, ε, στους πολίτες της Γερμανίας και αλλού. Η διαφάνεια είναι απαραίτητη και αυτή είναι η έκκλησή μου προς το Συμβούλιο και προς άλλους. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, είναι δύσκολη η καιρή, αλλά συμφωνώ απόλυτα με την θέση του κυρίου Ντεβίτε που λέει ότι λιγότερη δικαιοσύνη δεν είναι η σωστή λύση στην ε, οικονομική κρίση. Η έκκλησή μου προς το Συμβούλιο λοιπόν είναι να επιταχύνει τη διαδικασία. Ε, θα είναι απαραίτητο να συναντιόμαστε πάνω από δύο φορές κάθε εξάμεινο και σημαντικό είναι να συναντιόμαστε και με όλους τους παράγοντες που να μπορούν να ε, δώσουν ε, τεχνικές λύσεις στα θέματα που προκύπτουν. Αν αυτό γίνει είμαι βέβαιος ότι σε ένα χρόνο θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι τέτοιο, εάν υπάρχει πολιτική βούληση. Είναι σαφής λοιπόν η θέση του Κοινοβουλίου, η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσουν. Τώρα ήρθε η ώρα ε, να μετακινηθεί το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα. Ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές για την σημαντική συμβολή του, για τη βούλησή τους, ε, τη διάθεσή του, να παρευρεθούν εδώ, να μοιραστούν τι σκέψει του μαζί μα. Ε, ευχαριστώ όλου του ευρωβουλευτέ ε, και μπορώ να σα ανακοινώσω ότι θα συνεχίσουμε τι εργασίε τη επιτροπή ΛΥΜΠΕ στι 3 η ώρα το απόγευμα εδώ στην ίδια αίθουσα. Και να σα θυμίσω ότι το απόγευμα έχουμε ψηφοφορίε. Παρακαλώ θυμηθείτε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Σας ευχαριστώ όλους.